Colleagues, thank you for uh, being here this morning. Welcome to uh, today's committee meeting of security on security. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας είναι η έγκριση αυτής. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξή μας ο Δεν έχουμε βουλγαρικά, δανικά, εστονικά, φινλανδικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, λιθουανικά, λετονικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και σλοβενικά σήμερα. Δυστυχώς αυτό είναι το γλωσσικό μας καθεστώς, αλλά έχουμε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Η αυριανή μας συνεδρίαση θα αρχίσει 10 η ώρα και όχι 9. Παρόλο που θα χαιρόμασταν πολύ να σας δούμε στις 9 αύριο το πρωί, δεν θα έχουμε τίποτε να συζητήσουμε μέχρι τις 10. Οπότε, το πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξής μας, που είναι η δημόσια ακρόαση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και μελλοντικό στις αντίκτυπο στην ασφάλεια. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί. Εγώ την περιμένω με μεγάλη αγωνία. Είμαι σίγουρη ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι εδώ. Ο κύριος Τιμ Σουέιλς που είναι διευθυντής έρευνας στο Ίδρυμα Στρατηγικών Μελετών της Χάγης. Η κυρία Άντερσον που είναι εταίρος Έχουμε τον συνάδελφο Ντίκο, θα πω το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, τον ε, συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο τη Οκφόρδη και τον κύριο Ντίκοφ από το ε, τμήμα εξωτερικής πολιτικής και θεμάτων ασφαλείας. Η ακρόαση σκοπό έχει να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τη σχέση της με την άμυνα. Έχουμε ήδη συζητήσει εκτενώς ε, το θέμα των ε, drones και ε, των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, αλλά σήμερα θα συζητήσουμε κάποια ακόμη στοιχεία. Το πλήρω, δυναμικό, το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί, όμως έχει αρχίσει ήδη να εμφανίζεται στην, στις αγορές, όπως για παράδειγμα βλέπουμε με αυτοκίνητα και σε άλλους τομείς. Ε, έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι ε, προς πολύ καινοτόμες ε, εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. Φυσικά ένας από τους τομείς όπου θα γίνει αισθητό αυτό είναι η άμυνα. Τα αυτόνομα οπλικά συστήματα είναι ένα, ένας από τους τομείς, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της αναγνώρισης, επικοινωνίας, επιμελητία, ο σχεδιασμός ε, και ευρύτερα η, ε, η ανάπτυξη της στρατηγικής ε, ε, μακροπρόθεσμα. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχω τόσο εξέχουσε προσωπικότητε μαζί μου σήμερα για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δύο πάνελ θα έχουμε. Το πρώτο πάνελ θα μα κάνει μια ευρεία ε, επισκόπηση σε σχέση με το τι μπορούμε να περιμένουμε στον τομέα τη Άμυνα από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφους να κοιτάξουν μακριά στο μέλλον και να σκεφτούν ενδεχομένω και να υποθέσουν ποιε μπορεί να είναι οι μακροπρόθεσμε συνέπειε αυτή ε, της τεχνητής νοημοσύνης. Και στο δεύτερο πάνελ θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις προκλήσεις και ειδικότερα τις ρυθμιστικές προκλήσεις που θέτει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πολλά από αυτά τα ρυθμιστικά ζητήματα είναι βεβαίως οικουμενικής φύσεως και ισχύουν στη τεχνητή νοημοσύνη μη στρατιωτικής χρήσης και συνεπώς θα είναι ευρεία η εφαρμογή. Υπάρχουν όμως ανησυχίε όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στον στρατιωτικό τομέα και ελπίζω η Επιτροπή μας να ε, τα εξετάσει αυτά. Περιμένω λοιπόν εναγωνίω τι ε, σημερινέ συζητήσει, όπως είπα και στην αρχή. Και χωρί να καθυστερώ άλλο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Tim Schweiss, που είναι ο πρώτο ομιλητή του πάνελ μα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που οργανώνεται αυτή τη συζήτηση που είναι τόσο σημαντική και για την παγκόσμια ασφάλεια αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία εξέλιξη ε, στον γενικό τομέα που καλύπτεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, ε, ειδικότερα όσον αφορά την ε, αναγνώριση, υπάρχει τεράστια επένδυση, κυρίως από ιδιωτικούς εταίρους, από, τον ιδιωτικό τομέα, ε, με αύξηση της ισχύω και με αύξηση της διαθεσιμότητας μεγάλων συνόλων δεδομένων. Όπως είπε και η Πρόεδρος, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναστατώσει, θα μεταμορφώσει τη σχετική βιομηχανία, γιατί το βλέπουμε σήμερα και στα αυτοκίνητα που κινούνται μόνα τους, που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά πλησιάζει σιγά σιγά η στιγμή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις οικονομικές συναλλαγές, ε, βλέπουμε τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που γίνεται σε αυτό με το επίπεδο, σε αυτό με το επίπεδο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. πάρα πολλοί τομείς λοιπόν έχουν χαρακτηριστεί από αυτήν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ε, θα αλλάξει το είδος ή ο χαρακτήρας της σύγκρουσης, των συγκρούσεων στο μέλλον γιατί υπάρχει σχετική έρευνα και ανάπτυξη και στη Ρωσία και στις Ηνωμένε Πολιτείες ο στόχος είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της τρέχουσας γενεάς στρατιωτικών ικανοτήτων. Παράλληλα όμως σκοπό έχουν να ε, υπάρξει μια πρόοδος που μπορεί να δημιουργήσει και κάποια αναστάτωση. Επομένω, ο αντίκτυπο στην ασφάλεια τη τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια ανησυχία, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη μελλοντική ειρήνη και ασφάλεια. Θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια σε σχέση με το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν είναι, να ε, τονίσω κάποιε ε, παρεξηγήσει που μπορεί να υπάρχουν. Πρέπει να σκέφτεστε τη μελλοντική εξέλιξη τη τεχνητή ε, νοημοσύνη. Πέντε σημαντικά στοιχεία Πρώτον, ε, η σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα. Ε, είπα Ρωσία, Κίνα και θα αναφερθώ σε κάποιες εφαρμογές στην άμυνα της τεχνητής νοημοσύνης ε, σε αυτές τις χώρες και θα ολοκληρώσω με μία σύντομη αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να είμαστε ακόμη στην αύξουσα πλευρά του, ε, της τεχνητής νοημοσύνης, ε, όμως υπάρχουν ανησυχίες που δεν αδικαιολόγητε. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα σε σχέση με την πρόσφατη πρόοδο, για να είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποδείξει ότι μπορούν να υπερβούν την ανθρώπινη απόδοση, όσον αφορά, για παράδειγμα, την άμεση μετάφραση μπορεί για παράδειγμα να ε, αναγνωρίσουν ανθρώπινα πρόσωπα, να καταλάβουν τη διαφορά μιας ερώτησης από την κατάφαση. Ε, έχουν δημιουργήσει τα, νέα, τα δικά του συστήματα που μπορούν να αναγνωρίσουν κάποια ε, ασθένεια φυτική για παράδειγμα. Επίσης είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο πόκερ ή στο σκάκι για παράδειγμα. Ε, συνεπώς έχουμε ξεπεράσει τον, ε, την έννοια του Homo sapiens ε, ε, που είναι συνδεδεμένη με τη φυσική νοημοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναδυόμενη μορφή ευφυΐας και νοημοσύνης. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την άμυνα. Να σας πω τι ακριβώς εννοούμε. Δείξτε λίγη υπομονή, γιατί πρέπει να σας πω μερικά πράγματα για τον ορισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς, τι είναι η, η νοημοσύνη είναι το υπολογιστικό κομμάτι της ικανότητας να επιτύχει κανείς στόχους. Αυτός ο ορισμός αφορά εσωτερικές διαδικασίες, ε, ε, τους υπολογισμούς, την αυτοματοποίηση, τα εξωτερικά αποτελέσματα σε ένα περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ο ορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη φυσική και για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν δούμε ε, την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουμε ότι υπάρχουν ικανότητες που καλύπτουν καλύπτονται και από τη φυσική νοημοσύνη και που αφορούν για παράδειγμα του υπολογισμούς, τη δυνατότητα να σκεφτεί κανείς και να δράσει. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα λένε, λέγεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το να μπορούν οι υπολογιστέ να κάνουν κάτι που κανονικά χρειάζεται τη φυσική νοημοσύνη, όπω για παράδειγμα η συζήτηση, η λήψη αποφάσεων κλπ. Πρέπει να υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένα κομμάτια ε, που ε, θα βοηθήσουν την τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει αυτό. Αυτό ε, έχει άμεση σχέση δηλαδή με την εξέλιξη των μηχανών. Πρέπει να μπορούμε να καταλάβουν πολύ βασικές τάσεις και μεθοδολογίες, αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από διάφορες προσεγγίσεις στην εκμάθηση των μηχανών. Η Πρόεδρος ζητά ευγενικά από τον ομιλητή να μιλάει λίγο πιο αργά. θα... δεν χρειάζεται να σας ε, αναφέρω όλους αυτούς τους αλγορίθμους. Από τη στιγμή που είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη ε, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι ένας υπερ, υπερυπολογιστής που τα καταφέρνει όλα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές εφαρμογών ε, με, με, με διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν μια διάκριση που πρέπει να γίνει όταν σκεφτόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και τη μελλοντική πρόοδο στη τεχνητή νοημοσύνη. υπάρχει μια διάκριση μεταξύ της ε, πιο στενής νοημοσύνη τη γενική και υπέρνοημοσύνη. Ε, η στενή νοημοσύνη έχει να κάνει με τη νοημοσύνη των μηχανών, που σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τη νοημοσύνη των ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο, ε, για, μια συγκεκρι... για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το AlphaGo της Google, ε, υψηλή συχνότητας ε, συναλλαγές στο εμπόριο και εξειδικευμένα αυτοματοποιημένα συστήματα πέρα από την φυσική νοημοσύνη, ε, τα φίλτρα ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για παράδειγμα κάποια ε, στοιχεία που αφορούν το τα αντιβαλιστικά συστήματα. Τώρα ε, περνάμε στο επόμενο επίπεδο όταν οι μηχανές μπορούν να κάνουν όλες τις δραστηριότητες ε, ε, που μπορούν να κάνουν και οι άνθρωποι και μετά υπάρχει και η υπερνοημοσύνη και αυτό είναι η νοημοσύνη των μηχανών που υπερβαίνει την νοημοσύνη του ανθρώπου σε όλες τις δραστηριότητες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πλαισιώσουμε τη συζήτηση, καλό είναι να ξέρουμε ότι η στενή νοημοσύνη και οι σχετικές εφαρμογές... Ε, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να υπερβαίνουν τους ανθρώπους σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, αλλά είμαστε μακριά από μια κατάσταση κατά την οποία περνάμε στη γενική νοημοσύνη, στην υπερνοημοσύνη των μηχανών. Ένα κρίσιμο ζήτημα και ερώτημα αφορά την μελλοντική πρόοδο ε, στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ποιο σημείο θα περνάμε από το ένα επίπεδο στο άλλο δεν ε, συμφωνούμε ε, στα πάντα ε, ως προς αυτό. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Όμως υπάρχουν και εμπειρογνώμονες που θεωρούν ότι μπορεί να πάει πολύ γρήγορα. Ε, ας πούμε στο Google ε, υπάρχουν νέες εκτιμήσεις σε σχέση με το πότε θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο και ε, έχει αναθεωρηθεί αυτή η ημερομηνία από την Google στο 2029. Όσον αφορά τώρα τη γενική νοημοσύνη που ανέφερα προηγουμένως, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε ήδη να κάνουμε, μπορούμε ήδη να τα ενσωματώσουμε σε υφιστάμενες διαδικασίες και σε στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση. Και πολλοί αναλυτές, όπως και εγώ, θεωρούμε ότι θα συνεχίσει η εξέλιξη της στενής νοημοσύνης λόγω οικονομικών και πνευματικών επενδύσεων που αρχίζουν σιγά σιγά να υπάρχουν και από το δημόσιο και από το ιδιωτικό τομέα με επαναστατικές τεχνολογίες που σιγά σιγά θα είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμες. Άλλα πέντε σημαντικά σημεία που θα ήθελα να αποκομίσετε από τη σημερινή μου ομιλία αφορά τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας συγκεκριμένα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και η φυσική νοημοσύνη, η ανθρώπινη νοημοσύνη, δεν, είναι μια συγκεκρι... δεν αφορά μια συγκεκριμένη ικανότητα. Ε, μπορεί να συμπεριλάβει πολλές λειτουργίες σε πολλές εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση εικόνων, ήχων, ε, με γνώση, με επίλυση προβλημάτων, προγραμματισμό και όταν αφορά συνδυασμό με φυσικά αντικείμενα μπορεί να περάσει και στην εκτέλεση πολλών ε, δραστηριοτήτων. Ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά και για καλούς και για κακούς σκοπούς ε, στην άμυνα και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, η έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να είναι ευκολότερη σε περίπτωση μιας βίαιης σύγκρουσης και μπορούν ε, οι υπεύθυνοι λήψη αποφάσεων να περάσουν στην έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη, στην απορριζοσπαστικοποίηση ανθρώπων με πάρα πολύ ακραίες ιδέες, ε, μπορεί να βοηθήσει την διάσωση ζωών μέσω ιατρικής ιατρικής διάγνωσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει ώστε λιγότεροι άνθρωποι ε, να βρίσκονται στο πεδίο μάχης λόγω των μη επανδρομένων συστημάτων που αντικαθιστούν τα επανδρομένα. Επίση, μπορούν να κάνουν κάτι σε λεπτά όταν ε, μια ανθρώπινη ομάδα θα το έκανε σε μήνες. Μπορεί μια τεχνητή νοημοσύνη να, χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση μιας ε, αδυναμίας του αντιπάλου, να μπορέσει να αναγνωρίσει επιθετικά συστήματα με μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερο αυτοματισμό. Επίση, κάποιοι μπορεί, κάποια συστήματα επιθετικά μπορούν να ε, δώσουν σε μία μηχανή πλήρως τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάποια από τα ε, μειονεκτήματα και τα ευάλωτα σημεία του αντιπάλου και μάλιστα μπορούν να αντιδράσουν και πολύ πιο γρήγορα τα συστήματα αυτά. Η φυστάμενη γενεά λοιπόν αμυντικών ικανοτήτων μπορεί να χάσει την αξία της. Επίσης μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ε, ρήξη μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία, κάτι το οποίο φυσικά μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση μιας κρίσης. Ακριβώς επειδή η νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλούς και για κακούς σκοπούς, πρέπει να την προσεγγίσουμε με προσοχή και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων ε, εφαρμογών ε, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου του. Τρίτο σημείο, ε, αλγόριθμοι που βασίζονται σε λογισμικό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αλγορίθμους χρησιμοποιούνται με διτό τρόπο, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε στρατιωτικό και σε μη στρατιωτικό περιβάλλον. Επίσης μπορεί να γνωρίζετε το λογισμικό ε, έχει διάφορα επίπεδα, ε, δηλαδή υπάρχει ένας κωδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια μικρή παραλλαγή σε ένα άλλο σύστημα λογισμικού. Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που να μπορεί να δουλεύει με φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο και να την ε, προσεγγίσει, να την χρησιμοποιήσει σε κάτι ευρύτερο και γενικότερο. Είναι κάτι όμως το οποίο αν το χρησιμοποιήσει σε έναν άλλο τομέα μπορεί ξαφνικά να γίνει πάρα πολύ δαπανηρό. Όλες αυτές οι εφαρμογές λοιπόν έχουν διάφορα επίπεδα προσαρμογής. Το ζήτημα είναι η παραγωγή, η διασπορά όλων αυτών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορεί να ε, ελέγχεται σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει μια υποδομή ε, που αφορά για παράδειγμα τα οχήματα, ε, πολύ σημαντικές τεχνολογίες και μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που πρέπει να ελέγχεται. Ε, στον αμυντικό τομέα δεν ισχύει πάντοτε αυτό και αυτό περιπλέκεται ακόμη από το γεγονός ότι η έρευνα είναι από ιδιωτικού τομείς κατά μεγάλο ποσοστό που δεν είναι υπό τον κυβερνητικό έλεγχο ή δεν θέλουν να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ελέγξουμε την διασφάλιση και την παραγωγή αυτών των εφαρμογών. Αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί στο δεύτερο πάνελ. Πέμπτο σημείο, ε, η ε, τεχνητή νοημοσύνη, με τη στενή έννοια όπως ανέφερα, ε, υπάρχει περίπτωση να ε, επισπευθεί κατά την επόμενη ε, δεκαετία με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σημαντική για αμυντικούς οργανισμούς και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τον τρόπο με τον οποίο ε, αγωνίζονται, ε, μάχονται. Είναι λοιπόν προσαρμόσιμες αυτές ε, οι εφαρμογές, δεν είναι όμως ε, εύκολα ελεγχόμενες και μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση και να, οι συνέπειες αυτές να αυξάνονται συνεχώς. Φυσικά οι στρατιωτικοί οργανισμοί έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Οργανισμοί αμυντικοί, Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Κίνα παίρνουν την τεχνητή νοημοσύνη πολύ σοβαρά και περιμένω μια σοβαρή προσπάθεια να υπάρξει μια, ένα, μια συνέπεια αναστάτωση στον αμυντικό εξοπλισμό λόγω αυτού. Ε, γιατί υπάρχουν πολλέ τέτοιε μονάδε ε, στο Υπουργείο Άμυνα πολλών ε, των χωρών αυτών. Δεν μπορώ να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε. Ε, αλλά να σας ε, δώσω κάποια στοιχεία το 2014 οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ξεκίνησε μια στρατηγική με ειδικό στόχο διατήρησης της ε, στρατιωτική ε, ισχύω τη με αυτόνομα οπλικά συστήματα, προηγμένε, ομάδε ομάδες και προηγμένα άρματα μάχης. Ως τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας, πέρσι ξεκίνησε να λειτουργεί ένα κέντρο στρατηγικών ε, εφαρμογών με προπολογισμό 1,8 δις δολάρια. Ε, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, το οποίο θα έχει προπολογισμό 2,2 δις ε, δολάρια για να αρχίσει να αναπτύσσει περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στον αμυντικό τομέα. Ε, θεωρούν λοιπόν ότι όντως θα υπάρξουν εφαρμογές στο στρατιωτικό τομέα ε, και ε, ότι ο τομέας έρευνας και της ανάπτυξης σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του μέλλοντος. Και στην Κίνα υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση. Πέρσι είπε ότι θα είναι παγκόσμιος ηγέτης μέχρι το 2030. Ε, ο POA έχει σκοπό να περάσει από ε, να περάσει σε έναν ευφυή ε, πόλεμο έχει λοιπόν μία παδρομένα συστήματα, επιστημονικά συστήματα που τα μελετούν ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, ε, τεχνολογίας ε, και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν και για μη στρατιωτική χρήση να αναπτυχθούν αυτές οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Και η Ρωσία έχει σκοπό να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πούτιν είπε μάλιστα ότι όποιος είναι ηγέτης σε αυτόν τον τομέα θα είναι και ο ηγέτης του κόσμου. Υπάρχει το Ρωσικό Ίδρυμα Προηγμένης Έρευνας για να κλείσει το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και θέλει να καλύψει την καθυστέρηση στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων. Έχει θέσει το στόχο μάλιστα του 30% του στρατηγιωτικού εξοπλισμού που θα είναι ρομποτικός μέχρι το 2025. Η Ρωσία πολύ συχνά χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εστιασμένη σε αυτόνομα συστήματα για τις ΗΠΑ ε, και την Κίνα. Φαίνεται ότι ε, κυρίως βασίζεται στον κύκλο OODA Loop. Ε, η έρευνα και η ανάπτυξη αφορά κυρίως τα μοντέλα εγκαίρης προειδοποίησης, ε, συλλογή μυστικών υπηρεσιών, ε, ε, ανάλυση του πεδίου μάχης, ιατρική, ιατρικές διαγνώσεις, μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, μη επανδρομένα ή μη αυτόνομα συστήματα, νέα συστήματα διασποράς με αναλώσιμα οχήματα και τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να εξηγήσει τον εαυτό της ε, στους ανθρώπους για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι ακόμη και θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε. Προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει άμεση σχέση με ε, το πώς θα επηρεάσει αυτό την παγκόσμια ασφάλεια. Νωρί είναι ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει δείξει όλο τον αντίκτυπό τη. Θα ήθελα να σα πω όμω ότι υπάρχουν κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Θετικά στοιχεία. Θα υπάρχει καλύτερη στόχευση στην τεχνητή νομοσύνη και μπορεί να είναι πιο ανθρώπινος ο πόλεμος, για να το πω έτσι. Ε, δηλαδή είναι πιο εύκολο να υπάρχει να υπάρχουν καλύτερες ομάδες μάχης και λιγότερες ζωές ε, να ε, απειλούνται. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα και προηγουμένως, θα ανοίξει ευκαιρίες βελτίωσης της έγκαιρης προειδοποίησης ε, γιατί θα δώσει καλύτερες και πιο έγκαιρες πληροφορίες και μπορεί και να διευκολύνει την αποκλιμάκωση και στρατηγική διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, γιατί ε, μπορεί να διευκολύνει την ταχύτητα ε, λήψης αποφάσεων σε περιόδους κρίσεων. Αρνητικά στοιχεία τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλέ αρνητικέ συνέπειε επίση. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί σε χαρτοφυλάκια του στρατιωτικού τομέα όσο έχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να καταστήσει παροχημένα κάποια παραδοσιακά δόγματα και το πολιτικό κόστο του να μπει κανεί σε έναν πόλεμο μπορεί να είναι χαμηλότερο αν ε, λιγότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στο μέτωπο του πολέμου. Ε, και να γίνει αυτό πιο εύκολο δηλαδή. Ανώριμη τεχνητή νοημοσύνη στρατιωτικές πλατφόρμες μπορεί να οδηγήσει σε, μια, σε ανεξέλεγκτα αποτελέσματα, κάτι το οποίο συμβαίνει και στις οικονομικές συναλλαγές συχνά. Και κάτι ακόμη, η σύγκρουση μπορεί να επιταχυνθεί τόσο πολύ που η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει ε, ειδικότερα αν ο άνθρωπος δεν συμμετέχει καθόλου στη διαδικασία και οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο τεχνητή νοημοσύνης. Αυτό θα δώσει αντιπαλούς ένα βασικό δίλημα κατά πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να συμμετέχει και να υποστεί την ήττα ή αν θα συνεχίσει με την παρουσία του ανθρώπου ε, και να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ε, και ο χαρακτήρας και η φύση του πολέμου θα αλλάξουν συνεπώς δραστικά, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, ε, όπου ε, οι μηχανές θα πολεμούν η μία την άλλη. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία κυρίες και κύριοι για την ώρα, όμως το... τα σενάρια δείχνουν ότι υπάρχουν ε, ηθικά και νομικά ζητήματα που δεν πρέπει να απομονώνονται από τις στρατιωτικές και στρατηγικές ε, συνέπειες ε, της ανάπτυξης νέων στρατιωτικών τεχνολογιών. Αυτά από μένα σήμερα και θα περιμένω τις ερωτήσει και τα σχόλιά Σα Ευχαριστώ. Thank you very much for that. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πού βρισκόμαστε και το πού θα φτάσουμε όσον αφορά την ε, άμυνα στην τεχνητή νοημοσύνη και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Wendy Anderson, ε, η οποία όπως ε, είπα είναι ερευνήτρια στο κέντρο Νέας Αμερικανικής Ασφάλειας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγουμε καθαρά. Ευχαριστώ ε, πολύ ε, που συντονίζεται αυτό το ε, πάνελ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Φατίγκα, η οποία δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, όμως ελπίζω να συναντήσω κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Καθώς επίσης και την Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή ένα πιο σημαντικό θέμα γνωρίζοντας ότι όλοι έχουμε βέβαια ε, σημαντικά θέματα με τα, οποία, ε, τα οποία αντιμετωπίζουμε ανάλογα με τη χώρα από την οποία καταγόμαστε. Θα ήθελα όμως να πω ότι ευχαριστώ τα μέλη καθώς επίσης ε, και καλωσορίζω όλους σας ορισμένα γενικά στοιχεία. Ε, δεν είμαι μια ηγέτρια ε, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ασχολούμαι με το συγκεκριμένο τομέα εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω λέγοντας τι δεν είμαι. Είναι κάτι το οποίο κάνω από τα έξι όταν άρχισα να ε, την δεκαετία του 70 να διαλύω παιχνιδάκια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια εταιρεία και επίσης ε, ε, είμαι ερευνήτρια και στην ΣΥΝΑΣ και επίσης ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ασχολούμαι με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, με μια εταιρεία που ασχολείται με την άμυνα και την τεχνητή νοημοσύνη και εργάζεται για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επίσης και άλλες κυβερνήσει, και προσπαθούμε να βρούμε το πώς μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε ε, την τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα. Πρόσφατα είχα ε, την δυνατότητα να εργάζομαι ως υπεύθυνη προσωπικού ενό Υπουργού Εθνική Αμήνη των Ηνωμένων Πολιτειών ε, ήμασταν μαζί στο ε, Πεντάγωνο, ανεβήκαμε ε, τις διάφορες βαθμίδες, ε, μαζί με... Ακολουθούσα λοιπόν έναν υπουργό, ο οποίος ε, δεν ήταν μονάχα ένα σταθερό χέρι του Υπουργείου Αμήνης, αλλά ταυτόχρονα και ένας καινοτόμος όσον αφορά την ε, τον τομέα της άμυνας και εισήγαγε επίσης την εμπορική καινοτομία στην άμυνα των ΗΠΑ. Θα ήθελα να γνωρίζετε λοιπόν αυτό το πλαίσιο για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα την πηγή των σχολείων που θα κάνω σήμερα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας ε, λοιπόν νομίζω ότι έχουν υπάρξει μονάχα ελάχιστες ραγδαίες αλλαγές ε, στο πώς διεξάγεται πόλεμος. Ένας βασικός κατάλογος ε, θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή των όπλων, ε, τον, την αεροπορική υποστήριξη, τις ραδιοεπικοινωνίες, ε, την στρατηγική του Blitzkrieg στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την άφηξη των ε, πυρηνικών όπλων και θεωρώ λοιπόν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, βοήθησαν σε αυτές τις ε, σημαντικές αλλαγές και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε εν ώψη μιας ε, άλλης μεγάλης αλλαγής χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. και γνωρίζω ότι το, η υποεπιτροπή αυτή ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Ένα ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να σας θέσω εγώ είναι ποιος θα θέλατε να είναι ο ρόλος σας στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, χωρίς να περιλαμβάνουμε ίσως την παρούσα κυβέρνηση, ήμουν στην κυβέρνηση Ομπάμα, πολλοί από εμάς λοιπόν προσπαθήσαμε να θέσουμε αυτό το ερώτημα και τώρα το κάνω αυτό στο πλαίσιο της ε, ιδιωτικής βιομηχανίας αλλά και στο πλαίσιο μιας δεξαμενής σκέψης και διαφέρει από ό,τι όταν συμμετείχα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σας αφήνω λοιπόν με αυτό το ερώτημα έτσι για να αναλογιστείτε λιγάκι. Ε, ποιος θέλετε να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, όχι μονάχα των χωρών που εκπροσωπείτε ως ε, ευρωβουλευτές, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θέλετε να είναι ο ρόλος σας ε, και πιστεύω ότι μπορούν να δοθούν πολλές απαντήσεις. Έχω διαβάσει αρκετές ε, ενδιαφέρουσες απαντήσεις πάνω σε αυτό το ερώτημα μέχρι στιγμής, όμως θα ήθελα μακροπρόθεσμα να μάθω τις ε, ιδέες σας, ε, τις συστάσεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να έχετε κάποιον Αμερικανό να σας έρχεται και να σας λέει τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Όμως ως σύμμαχος ε, και αντιλαμβανόμενοι το ρόλο μου και, τις, ε, ε, και του κοινού τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τα προβλήματα, το λέω αυτό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να αποδεχτώ τον, τους ορισμούς που έδωσε ο Τιμ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι είχε έναν πολύ ωραίο τρόπο όχι μόνο για να μιλήσει το πόσο ευρύ είναι αυτή η όρη αλλά έγινε και πολύ καλή δουλειά κάνοντας αυτή την ε, διαφοροποίηση μεταξύ των τριών ειδών τεχνητής νοημοσύνης. Θα αφήσω λοιπόν τους ορισμούς που χρησιμοποίησε και θα τους αποδεκτώ και θα πω ότι συμφωνώ με την ορολογία την οποία παρουσίασε και θα την υιοθετήσω και στα δικά μου σχόλια. Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάποιος που έρχεται τώρα στη συζήτηση ίσως να πιστεύει κάτι τέτοιο όμως ε, γνωρίζουμε την συνεισφορά του Alan Turning, ε, γνωρίζουμε όλα τα κεφάλαια τα τελευταία 30 με 60 χρόνια και τις ε, αλλαγές που έγιναν στην, στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, όμως πιστεύω ότι θα βοηθήσει ε, η συζήτηση. Ίσως τα απομακρυσμένα κινούμενα τα κινούμενα εξ αποστάσεως αυτοκίνητα ίσως να μην βοηθούν, τα, ε, τα αεροπλάνα μπορούν εξ αποστάσεως να τα χειριστούν και να στοχεύσουν συγκεκριμένους ε, στόχους. Έχουμε τα ημιαυτόνομα σύστημα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στα πεδία μάχης. Μπορώ να σας σκοτώσω από βαρεμάρα λέγοντας ε, τα όσα χρησιμοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείε όλα αυτά τα μη αυτόνομα συστήματα, όμως ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ σήμερα στα σχόλιά μου ότι αυτό το οποίο μας περιμένει είναι τεχνολογίες οι οποίες μαθαίνουν στην πορεία. Ε, υπάρχουν ε, αλγόριθμοι, ε, όμως ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις δικές τους πληροφορίες και κατευθυντήριες δράσεις με βάση τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν, οι οποίες ίσως να μην ήταν αρχικά προβλέψιμες. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα περιγραφή που δείχνει αυτήν την τρομερή αλλαγή μελοδραματικό ίσως να ακούγεται, όμως ταιριάζει σε αυτό ε, το πλαίσιο. Διότι το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεκινήσει την πορεία του. Την πορεία του. Ήδη βρισκόμαστε σε έναν αγώνα όπλων, δεν θα ήθελα να το πω έτσι ακριβώς, διότι δείχνει ε, μια ανταγωνιστικότητα ε, και δείχνει το ποιος θα ξεπεράσει ποιον. Νομίζω λοιπόν ότι το ενδιαφέρον όσον αφορά την εισαγωγή της ε, τεχνητής νοημοσύνης ε, θα αποτελέσει μια σημαντική γεωπολιτική διαφοροποίηση και ταυτόχρονα έχει να κάνει με το πώς θα αναπτύξουμε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ε, και μακροπρόθεσμες ε, ε, ημερήσεις διατάξεις, σχέδια σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η γραφειοκρατία σας και μας έχουν μία κάποια φήμη και είναι ενοχλητικό διότι συνεχώς θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε τις αναγκαίες παρακάμψεις ε, για να εισάγουμε την αναγκαία καινοτομία ιδιαίτερο ε, στον ε, χώρο της άμυνας. Ο κόσμος φυσικά και έχει κάποιες ανησυχίες, σκέφτεται ίσως τον εξολοθρευτή, όμως ίσως η ως γνωρίζοντες να το καταλαβαίνουν αυτό. Όμως βρισκόμαστε ακόμα στα σπάργανα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να ξεκινήσουμε αμέσως. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τις ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, τα, τις ηθικές συνέπειες ε, ε, και όλα αυτά. Όμως αυτός ο ενθουσιασμός που υπάρχει όσον αφορά τα ρομπότ που σκοτώνουν από αμερικανικής σκοπιάς και από κάποιον ο οποίος περνάει πολύ χρόνο στην Silicon Valley είναι πολύ πρόωρο αυτό το άγχος Οπότε αυτό ας είναι στο τέλος του καταλόγου, απέχουμε δεκαετίες ακόμα. Όποιος θέλει βέβαια μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου. Ε, Τώρα το που βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πίσω ε, σε αυτόν τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης ε, και μπορώ να αναλύσω στη συνέχεια ε, το επιχείρημα αυτό. Δεν είναι απεσιοδοξία, απλά εξετάζω πώς είναι η χρηματοδότηση, η δεξαμενή ταλέντων, το πώς έχει η κατάσταση. Και όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνω στην ανάλυση μου και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε πίσω σε σχέση ας πούμε με την Κίνα. Ήθελα να επικεντρωθώ στις ε, παρατηρήσεις μου και τις ε, συστάσεις μου προς αυτό το κοινό οτι όλοι σιγά σιγά αρχίζετε να σκέφτεστε το πώς θα λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι περιγράφοντας <coughs> τις Ηνωμένε Πολιτείε και ισχύει και στην Ευρώπη ότι αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις ε, της τεχνητής νοημοσύνης στην μηχανική μάθηση σε ε, επίπεδο ε, εμπορικό αλλά και στρατιωτικό τα τελευταία χρόνια είχα 20-30 συζητήσεις ε, και αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αλλά και πολιτικοί και ευρωβουλευτές ε, συζητούν τις επιρροές που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην συμμαχία και στις στρατιωτικές δυνατότητες της συμμαχίας, καθώς επίσης ε, και γενικότερα στις επιρροές της τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Και φαίνεται ότι είναι μια ε, συζήτηση που έχει δύο μέρη. Από τη μία έχουμε τους ε, πολιτικούς των ΗΠΑ που δεν εποφελούνται την των δυνατοτήτων της ε, τεχνητής ε, νοημοσύνης ε. και πιστεύω ότι αυτό θα είναι σημαντικό και για άλλες αποφάσεις που θα είναι ε, ληφθούν. Η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο και έχει περιγραφεί πολύ συχνά στο να ε, χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους τα προσωπικά σας ε, δεδομένα. Δεν ε, είναι ενθουσιασμένος όλες οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, ο Μακρόν από την Γαλλία έχει διαφορετική στάση στην, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Όμως ας σκεφτούμε την ε, Γαλλία ως ε, μια startup. Είναι ε, κάτι ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να προκύψει από αυτή την χώρα και κάτι πολύ αισιόδοξο το οποίο μπορεί να δηλώσει ένας ηγέτης ευρωπαϊκής χώρας. Ήταν πολύ ωραίος τρόπος να το θέσει. Πώς γίνεσαι μια startup χώρα όσον αφορά την ε, τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Θα τελειώσω όμως ε, λέγοντας, ε, αναφέροντας έξι πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν ακόμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετάσχουν στην, Ευρωπαϊκή, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορούν οι σύμμαχοι να καλύψουν το χάσμα διαλειτουργικότητας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έξι πράγματα λοιπόν. Πρώτον, μην περιμένετε. Δεν προσπαθώ να σας πατρονάρω. Βρισκόμαστε και εμείς στο ίδιο σημείο για διαφορετικούς, διαφορετικούς λόγους. Το τρένο έχει ξεκινήσει και πλέον ε, θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με τα σοβαρά ερωτήματα. Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά ε, το αγοράζω Αμερική δεν είναι ε, μονάχα μια αμερικανική τεχνική πώληση προϊόντων μας. Τρίτον, η ε, τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ε, προσέγγιση από όλη την κυβέρνηση. Τέταρτον, είναι ίσως πειρασμός να προστατεύσουμε την την ε, βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη εμποδίζοντας ε, την ε, αμερικανική βιομηχανία, όμως το κλειδί είναι η συνεργασία. Και εμείς όμως δεν είμαστε τέλειοι, όμως θα πρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί στον ανταγωνισμό. Πέμπτον, προφανώς το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα δύο βασικότερα κομμάτια του παζλ ε, τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη ε, και το πώς ε, όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και έκτον ο καθορισμός των κανόνων. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό δεν μπορούμε να κάτσουμε στην άκρη και να περιμένουμε ότι απλά θα ακούσουμε, θα ακουστούν, θα γίνουν ακουστές οι ανησυχίε μας και ότι απλά θα περιμένουμε να ε, λυθεί το πρόβλημα μόνο του. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε για τις χώρες μας και την άμυνα τους, αλλά και για τη συλλογική μας άμυνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις προκλήσεις που μας θέσατε. Αυτός είναι και ο ρόλος μας για το μέλλον. Ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές για τις πολύ ενημερωτικέ εισηγήσει. Αρχίζουμε τώρα το διάλογο. Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. δεν ε, διασκεδάστηκαν οι ψυχίες μου. Αν λέτε μάλιστα ότι θα πρέπει να αναρτηθούμε το δικό μας ρόλο. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό στο Κοινοβούλιο. Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει απαγόρευση διεθνή για αυτά τα όπλα. Και πρόσφατα είχαμε και ένα ψήφισμα όπου 566 βουλευτές υπερψήφισαν επειδή φοβάστε ότι περνάει ο χρόνος και θέλουμε η Κομισιόν και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν μια θέση γιατί αν πάμε στον ΟΗΕ με κάτι συγκεκριμένο πρέπει να έχουμε μια θέση πρώτα. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν. Και θα πρέπει πραγματικά η Ευρώπη να απαγορεύσει αυτά τα όπλα. Δεν μένουν δεν είναι θέμα μάλλον δεκαετιών ή αυτής δεκαετίας, των επόμενων δύο δεκαετιών. Θα πρέπει να έχουμε ένα τα αιώνα. Θα πρέπει να σταματήσουν λοιπόν τα όπλα αυτά με μια διεθνή απαγόρευση. Και ακούγοντά σα, κύριε Άντερσον, φαίνεται ότι ο αγώνα στον εξοπλισμό συνεχίζεται. Εμεί είμαστε πίσω, έχουμε μείνει πίσω. μπορεί θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά. Συνεργασία την Ευρώπη κλπ. Αλλά μπορούμε να τα σταματήσουμε αυτά. Γιατί ανησυχώ πραγματικά. Ίσως το επόμενο πάνελ που θα μιλήσει για τι αποφάσει να το σχολιάσει, αλλά δυστυχώ πρέπει να φύγω. Για τη λήψη αποφάσεων λοιπόν, για την ευθύνη. Ποιο είναι υπεύθυνο. Ποιον θα εγκαλέσουμε αν κάτι πάει στραβά ή αν πέσουν αυτά τα οπλικά συστήματα στα λάθος χέρια. Γιατί μπορεί να συμβεί και το ξέρουμε. Αν είμαστε δημοκρατίες με δημοκρατίες που λειτουργούν τώρα, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι πολιτεύματα θα έχουμε και τι θα αλλάξει και πώς θα προσπαθήσουμε αυτά τα οπλικά συστήματα. Οπότε ανησυχώ πάρα πολύ και ανησυχώ περισσότερο μετά τη δική σας την εισήγηση. Σαμκέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να θίξω ένα άλλο θέμα εγώ. αυτό που ακούσαμε προηγουμένως νομίζω ισχύει ότι δηλαδή αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να σταματήσει. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να θίξω κάτι διαφορετικό. Η κούρσα στα τεχνολογικά όπλα μέχρι τώρα πώς ήταν. Είχαμε ας πούμε κάποιες έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές, GPS, ε, υπολογιστές κτλ. Και, και η στρατιωτική χρήση ήταν πάντα πρώτη. Και μετά σιγά σιγά αυτές οι στρατιωτικές χρήσεις έφτασαν και στους πολίτες. Σήμερα όμως αντιμετωπίζουμε μια τελείως νέα κατάσταση. Οπότε έχω την εξής ερώτηση. Μιλάμε για την έρευνα για τεχνητή νοημοσύνη που διεξάγεται όμως σε διάφορους τόπους, σε διάφορα μέρη. μπορούμε να έχουμε έτσι μια ταυτόχρονη εξέλιξη πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Η αυστηρά, η καθαρά στρατιωτική έρευνα αφορά προφανώς το στρατό και η πολιτική χρήση δεν εφάπτεται αυτή τη στρατιωτική χρήση. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να έχουμε μια διπλή διτή χρήση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τον έλεγχο, γιατί θα πρέπει να, χρησιμοποιήσουμε έλεγχο για αυτές τις εφαρμογές. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλής, ευχαριστώ πολύ. Είδα ένα άρθρο στον New Yorker πρόσφατα, το Μάιο ήταν φέτος, που ρωτούσε πόσο θα έπρεπε να μας φοβίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ted Friend το έγραψε που μοιάζει πολύ με το δικό μου το επώνυμο. Αλλά εδώ ακριβώς τελειώνει η καθεομοιότητα. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι έγραφε, αλλά τέλος πάντων να παραθέσω μια σύντομη παράγραφα από αυτά που έγραψε, που είπε ότι ακριβώς πώς και πότε η περιέργεια μας θα μας σκοτώνει. Γιατί είμαστε περίεργοι. Φοβούνται οι μηχανικοί και οι επιστήμονε ότι από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε δομές τεχνητής νοημοσύνης θα έρθει η καταστροφή. Ο Έλον Μάσκ που γνωρίζουμε όλοι με την Τέσλα κτλ. προέβλεψε μια δικτατορία ανήθικη από την οποία δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε εύκολα. Ο Στίβεν Χόκκιν είχε πει ότι η τεχνητή νομοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην, στο τέρμα, στο τέλος της ανθρώπινης ράτσας, των ανθρωπινών όντων. Οπότε μήπως θα έπρεπε λοιπόν να πάμε πιο σιγά στην τεχνητή νοημοσύνη ή αντίθετα θα έχουμε μια προσέγγιση Godzilla καταστροφής τεράστια δηλαδή που θα μετουσιωθεί σε ένα είδος ε, ρομπότ τεράστιου που θα μας δυναστεύει. Θα ήθελα την άποψή σας από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τελευταία ερώτηση. Ήταν αυτή. Και μετά θα ζητήσω από τους δύο να απαντήσουν. Κύριε Άντερσον πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ να σας απαντήσω και εκτιμώ το πάθος και την ειλικρινιά σας με τα οποία διατυπώσατε το ερώτημα. Τα σημεία κινησή μας μπορεί να διαφέρουν και αυτό οφείλεται βεβαίω στην ιστορία μας και στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων θα σας δώσω τη δική μου άποψη. Δεν λέω ότι είναι απόλυτη αλήθεια, αλλά είναι προσωπική μου άποψη που έχει σφυρλατηθεί τέλο πάντων όλα αυτά τα χρόνια που όπου εργάστηκα στο τομέα της άμυνας στη ΣΥΠΑ τόσα χρόνια. Ελπίζω μη μακάρι να ζούσαμε σε ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά, χωρίς άλλα προβλήματα. Εύχομαι να υπήρχαν πολλά που δεν είναι όμως έτσι. Εύχομαι τα πράγματα να ήταν όπως λέτε εσείς. Γιατί δεν πιστεύω στο θα έπρεπε ή στα θα έπρεπε βάσει δική μου εμπειρία, βάσει μου πορεία. Γιατί δεν έχουν τα θα έπρεπε σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε, αν δούμε τι αναλογίες, και παρά το γεγονό ότι πολλέ χώρε έχουν υπογράψει τη συνθήκη απαγόρευση ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, αυτό δεν απέτρεψε την Βόρεια Κορέα από το να δημιουργήσει πυρηνικό οπλοστάσιο κλπ. Έχουμε κάποιο οπλοστάσιο αποτροπή. Οπότε, κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή λάθο, Εγώ είμαι ένα από αυτούς Αμερικανού που δεν χρειάζεται να έχουν δίκιο, απλά και μόνο σα λένε την άποψή του. Εδώ έχουμε να κάνουμε τη δυνατότητα αποτροπής στην τεχνητή νομοσύνη. Γιατί πολλές άλλες ε, τεχνολογίες ήταν αρνητικές. Κάποιες τεχνολογίες δεν είναι αποτελεσματικέ και δεν έχουν και λόγο ύπαρξη. Και θα ήθελα να, να κάτι που είπε ο κύριος Φρόιντ για τον Elon Musk που έλεγε ότι η τεχνητή νομοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στον όλεθρο κλπ ειλικρινά να σας πω ότι η τεχνολογία από μόνη της, από τη φύση της, είναι ουδέτερη. Δεν είναι έμφυτα καλή ή κακή. Οι άνθρωποι την κάνουν αυτό που είναι. Οπότε, σε υπεύθυνα χέρια μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη ικανότητα για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Κάθε σύγχρονη ή μεταμοντέρνα τέλο πάντων φάση της εποχής που ζούμε καθορίζεται από κάποια μορφή δημιουργικότητας ή κάποια δυνατότητα επινόησης που ξεκλειδώνει το δυναμικό της τεχνολογίας. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Δεν πιστεύω απαραίτητα ότι πάντοτε ε, είναι θετικό αυτό, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια ε, Αμερική εμείς μάλλον μπορούμε να αποδείξουμε ότι πάνε σχετικά καλά τα πράγματα, αλλά από μόνη της τεχνολογία είναι ουδέτερη. Μπορεί να είναι θετική λοιπόν, μπορεί να είναι και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά καταλαβαίνω τις αμφιβολίες και τους δισταγμούς που αναφέρετε, αλλά θεωρώ ότι πια αυτή η κατάσταση είναι μη ε, μετατρέψιμη. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε, να αποκλείσουμε την ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη και απλά και μόνο καθίστε να παρακολουθήσετε τι κάνουν οι Κινέζοι, α πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, πρέπει να δούμε κατά πόσο θα έχουμε επενδύσει ε, ή δισεκατομμύρια που επενδύονται στην ε, Σαγκάη ή άλλα προγράμματα με τεράστια κονδύλια κτλ. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά υπάρχουν αμφιβολίες, είναι αλήθεια. Αλλά αυτά που σας λέω βασίζονται στα γεωπολιτικά δεδομένα τεχνολογικών επενδύσεων σε όλο τον κόσμο. Παγκοσμίω και οι Κινέζοι, σύμφωνα με τον Eric Σμιτ, που ήταν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος στην Alpha Group, την μητρική εταιρεία της Google, ο κύριος Σμιτ ε, του είπαμε πρόσφατα ότι κύριε Σμιτ, αν θα μας λέγατε σήμερα πόσο καιρό θα χρειαστούμε μέχρι οι Κινέζοι πραγματικά να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Μας είπε 4-5 χρόνια θα χρειαστούν για να τι ξεπεράσουν τις ΗΠΑ Μπορεί να κάνει λάθος, αλλά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η τάση προ τα εκεί πάει. Οπότε θα ήθελα να πω ότι σήμερα αυτές οι ειλικρινείς και δυστυχώς υποχρεωτικά ατελείς ανταλλαγές είναι χρήσιμες όπως εδώ σε αυτό το φόρουμ. Τώρα θα πρέπει να δαπανίσουμε χρόνο για να συζητήσουμε ακριβώς πώς θα αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε την τεχνολογία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς δεν θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε να τα έχουμε κατά νου όλα αυτά, αλλά νομίζω θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα απαγορεύσης γιατί νομίζω μια απαγόρευση ακριβώς δεν θα αποτρέψει την πρόθεση η οποία διέπει την τεχνολογία, η τεχνολογία της χρήσης και θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το συστηματικό το οποίο θα, ταυτόχρονα όμως δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και θα προστατεύει και τις χώρες μας, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη κτλ. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που είπατε και πάλι και πραγματικά ε, εκτιμώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και Πρόεδρος. Και τώρα για απαντήσεις και συμπεράσματα ο άλλος ηγητής μας. Κύριε θα θα και το πολύ σημαντικό. Αν δούμε τη στρατιωτική ιστορία, νομίζω ότι ποτέ δεν είχαμε μια κατάσταση όπου οι χώρες, τα κράτη δεν εποφελήθηκαν της ευκαιρία να ξεπεράσουν τεχνολογικά τους ανταγωνιστές τους. Αν δούμε, ας πούμε, τα αριοθούμενα ή τους πυράβλους, τη στρατηγική τους χρήση ή τον πόλεμο των ε, υποβρυχίων, τα τάγκς ε, σε αντίθεση με τα άλογα κτλ. Πάντοτε τα κράτη υιοθετούσαν την τεχνολογία η οποία σε επέτρεπε να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές. Και αυτό έμαθα μελετώντας, σπουδάζοντας τον πόλεμο. Τούτου λεχθέντος, αυτό σημαίνει ότι αν εμείς ως Ευρωπαίοι θέλουμε να επηρεάσουμε την ανάπτυξη τεχνολογίας στο μέλλον, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται, θα πρέπει να έχουμε μια βάση γνώσης, αλλά θα πρέπει επίσης να εμπλακούμε, να συμμετάσχουμε, ώστε να καθορίσουμε τις προδιαγραφές, τα πρότυπα. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσει και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να προωθήσουν τα πρότυπά μα και τις προδιαγραφέ μα και βέβαια η, δεύτερη συνεδρία γι' αυτό θα μιλήσει και αυτό αφορά και την διτή χρήση της τεχνολογίας στην οποία αναφερθήκατε γιατί δεν έχουν όλες τις τεχνολογίες διτή χρήση γιατί στο πεδίο της στρατιωτικής χρήσης τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα. Το περιβάλλον είναι κάπως ιδιαίτερο. Ε, ίσως λοιπόν χρειαζόμαστε και καλύτερα συστήματα, αλλά ακριβώς για να θέσουμε αυτά τα πρότυπα και να αποτρέψουμε την αυθαίρετη χρήση τους, νομίζω θα πρέπει να εμπλακούν και να συμμετέχουν οι κυβερνήσεις. Και τρίτον, σε σχέση με αυτό το θαυμάσιο άρθρο στον New που και εγώ διάβασα είναι σημαντική αυτή η άξιση, είναι γεωμετρική αυτή η πρόοδος, είναι αριθμητική αυτή η πρόοδος, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα ήθελα να θίξω το γεγονός ότι η δεκαετία του 90 είχαμε την εμφάνιση του ίντερνετ και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού άρχισαν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και νομίζω κάπου εκεί στο 2006 ο Bill Gates ένας άλλος οραματιστής είπε ότι η τεχνολογία της πληροφορικής θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στο άμεσο μέλλον σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή το email, ε, οι αγορές online κτλ. Τι έχει μεσολαβήσει λοιπόν από το 6 μέχρι το 18 σήμερα. Είχαμε το YouTube, το WhatsApp, τα κοινωνικά δίκτυα και ο αντίκτυπό του στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να σας πω, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι αυτές οι πρόοδοι οδήγησαν σε ποιοτικέ πρόοδου. Ήταν αριθμητικέ πρόοδοι που οδήγησαν σε ποιοτικέ πρόοδου. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τελειώσατε, αλλά έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε ότι οι νέες τεχνολογίες είναι ουδέτερες. Εγώ διαφωνώ. Εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός ο ίδιος και δεν το θεωρώ αυτό ουδέτερο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια αξιολόγηση των κινδύνων αυτής της τεχνολογίας. Βεβαίως θα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα. Αυτό είναι αναφεσβήτητο αλλά δεν είναι στην ουσία δικιά μας δουλειά, όπως είπατε και εσείς, να εξετάσουμε τους κινδύνους και να βρούμε να αναπτύξουμε λύσεις οι οποίες ακριβώς αποτρέπουν ή εξωτερών τους κινδύνους. Είναι αλήθεια ότι η Κίνα έχει προχωρήσει πολύ. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς από τη μεριά μας ότι θα κάνουμε τα ίδια. Η δικιά μας η απάντηση πρέπει να συνίσταται στο πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, πώς θα έχουμε αυτές τις συνθήκες, πριν επεκταθούν παγκοσμίε αυτές οι τεχνολογίες. Και η αλήθεια είναι ότι η συνθήκη της μη διάδοσης έλαβε χώρα αργά, καθυστερημένα. Αν είχε γίνει νωρίτερα θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ακόμα χρόνο, όχι πολύ, και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και αυτή είναι η δική μου άποψη προσωπική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό μας πηγαίνει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την ε, νομοθεσία και την έγκαιρη αντιμετώπιση της. Ναι, να σχολιάσω κάτι άλλο. Ως φυσικός ξέρετε για το Manhattan Project, ξέρετε για το ποιοι ε, επιστήμονες συμμετείχαν και τι σκέφτηκαν στο τέλος, τι άποψη είχαν. Αυτό όμως δεν τους απέτρεψε από το να φτιάξουν την πυρηνική βόμβα. Και η ΕΠΑ και η Σοβιετική Ένωση χρειάστηκε να επινοήσουν διάφορους τρόπους ελέγχου να παληθεύσεις ελέγχους και το οποίο θα συζητήσουμε μετά ώστε να επιβλέπει ο ένας, τον άλλο, ο ένας του άλλου τις πυρηνικές το πυρηνικό πλαστάσιο ώστε να μην έχουμε ακριβώς εξοπλισμό, ε, κούρσα για πυρηνικό εξοπλισμό οπότε πρέπει να δούμε ακριβώς τι τρόπους τεχνολογικής επαλήθευσης θα μπορούσαμε να έχουμε σε ένα πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά το αφήνω αυτό για το επόμενο πάνελ το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ναι, ναι, πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά. Ωραία το πάτε και σχεδόν με κάνατε περιττή. Αχρίαστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Συνάδελφοι, τώρα είναι πραγματικά στιγμή να πάμε στα πιο λεπτομερή ζητήματα σε σχέση με την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε σχέση με το τομέα της άμυνας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεφό. Είναι από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρωπότητας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η τεχνητή λοιπόν νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο και το ΜΜΕ και αλλού και μεγάλο από αυτό το ενδιαφέρον καθοδηγείται από μια παρανόηση και από μια υπερβολή. Αλλά θα είναι σημαντική η τεχνολογία η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό βέβαια είναι γνωστό, αλλά το πώς θα εξελιχθεί θα καθορίσει τον 21ο αιώνα. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και υπέρ και κατά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε καταρχάς τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπαμε προηγουμένω, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια γενικού σκοπού τεχνολογία που συνδέει τεχνολογίες, ε, μεσοδική κάψη, ηλεκτρικό ρεύμα, μικροεπικραστές κτλ. Όπου μεταμορφώνουμε κάποιες ιστροές σε διάφορους τομείς, ενέργεια, μεταφορές κτλ. Κάνοντας το αυτό, έχουμε κάποιες επιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα μεταμορφώνουμε την κοινωνία, την οικονομία και το στρατιωτικό τομέα. Είναι δύσκολο να λέξουμε κάποιες τεχνολογίες όπως είπαμε επειδή έχουν τόσο βαθιά τη χρήση και έχουν διαχυθεί στην οικονομία. Τέλος, ο αντίκτυπος των γενικών τεχνολογιών είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα σα αναφέρω ότι η τεχνητή νοημοσία, ε, η νοημοσύνη συγγνώμη, ε, θα είναι αυτή που θα επιφέρει τι μεγαλύτερε μετατροπέ, μεγαλύτερε μεταμορφώσει. Και νομίζουμε, θεωρούμε ότι υπό τη σημερινή τη μορφή, χωρί άλλε αλλαγέ, μπορεί ήδη από μόνη τη να αλλάξει παγκοσμίω τα δεδομένα. Και παρόλο που θα μπορούσε να σταματήσει θα μπορούσε να σταματήσει η ανάπτυξη τη ε, τεχνητή νομοσύνη σήμερα, θα μπορούσε να, να έχει μεγάλε επιπτώσει στην ανάπτυξή τη στο άμεσο μέλλον. Αυτά θα μπορούσαν βέβαια να οδηγήσουν σε αύξηση της των ανισοτήτων, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, μεταφορά εξουσίας, ε, έλλειψη σταθερότητας και ασφάλειας πυρηνικής, επιτός στην οικονομία και όπως συζητάμε σήμερα την στρατιωτικοποίηση της θεμητής νομοσύνης. Παρ' όλα αυτά, η πρόοδος δεν έχει σταματήσει. Προχωράει η πρόοδος της νομοσύνης κάθε χρόνο. Βλέπουμε ε, στο τομέα της γνώσης, στο σχεδιασμό, στην ε, πραγματογνωσύνη και στη σκέψη για το μέλλον της νοημοσύνης. Είναι δύσκολο λοιπόν να προβλέψουμε τις προκλήσεις και τη χρήση που θα ανακύψουν τα επόμενα 20 χρόνια, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γίνει με τις ριζικές μετατροπές ή τις αλλαγές στην ανθρώπινη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι τις απαντήσεις αυτές δεν τις ξέρουμε. Και όποιος κάνει προβλέψεις, είτε ξέρουν κάτι που δεν μας λένε, είτε κάνουν λάθος στις προβλέψεις τους. Εδώ σας έχω ένα γράφημα για τις πεπιθήσεις των ερευνητών το 2016 για πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Έχουμε εδώ διάφορους μεταβλητές που λάμβανε υπόψη το πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ θα δείτε λοιπόν ότι με ένα δηματολόγιο απαντήσεων υπάρχει απόκληση απόψεων. Κάποιοι δίνουν μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουμε δραστικά σε 10 χρόνια. Άλλοι δίνουν χαμηλή ε, και λένε, πιθανότητα και λένε σε 100 χρόνια και οι περισσότεροι είναι κάπου ανάμεσα. Αν λάβουμε λοιπόν τον μέσο όρο, καταλήγουμε στο ίδιο που λέει στην ουσία ότι κάποια στιγμή τα επόμενα 10-20 χρόνια όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά ούτε για τα επόμενα 100 ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία. Υπάρχουν διάφορες ε, πτυχές της τεχνητής νομοσύνης που θέτουν προκλήσεις για τις, ε, για τις κυβερνήσεις. Είναι γενικού σκοπού τεχνολογία, οπότε μπορεί να επιφέρει μεταμορφώσεις, μετατροπές και είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο. Τα υπέρ και τα κατά ε, μπορεί να διαχυθούν. Μπορεί να αφορούν, ας πούμε, περιφέρειες, κράτη, επιχειρήσεις, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Οπότε έχουν, λοιπόν, έχουμε λοιπόν προκλήσεις οι οποίες είναι παγκόσμιες, οπότε χρειάζεται παγκόσμια πρόκληση για να αντιμετωπιστούν. Πάντως θεωρώ ότι η πηγή για τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ακριβώς το πώς συμμετέχουν οι διάφορες ισχυρές χώρες σε αυτόν τον αγώνα, της, σε αυτή την κούρσα της τεχνητής ε, νοημοσύνης. Υπάρχει σύγχυση σε σχέση με τις κούρσες για την τεχνητή νοημοσύνη και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ας διαχωρίσουμε καταρχάς για τις διάφορες δυναμικές που υπάρχουν. Κάποιες οι οποίες έχουν ονομαστεί κούρσα εξοπλισμού, αλλά όχι μόνο. Καταρχάς ο ανταγωνισμός. Έχουμε τους ερευνητές που προσλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, οι βέβαια ταυτόχρονα διαμαρτύρονται για το πόσο ακριβό είναι να προσλάβουν ταλέντα από τη Silicon Valley. Έχουμε καταρχάς λοιπόν αυτό το είδος κούρσας ανταγωνισμού, όπου υπάρχει τέλο πάντων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Αλλά αυτό δεν αφορά άμεσα την, ε, το στρατιωτικό σκέλος, γιατί ωφελεί κατά κάποιο τρόπο την κοινωνία. Μετά έχουμε το μη στρατηγικό οικονομικό ανταγωνισμό. Και πάλι εδώ η μεταφορά αυτή τη κούρσα δεν είναι σωστή. Δηλαδή ο οικονομικό ανταγωνισμό είναι στρατηγικό ανταγωνισμό. Ο οικονομικό ανταγωνισμό είναι ωφέλιμο, ενώ ο, η κούρσα ανταγωνισμού δεν είναι. Και επίση χρειαζόμαστε συχνά μια εθνική στρατηγική χωρί ανταγωνιστικέ επενδύσει στην εκπαίδευση, α πούμε, στην άμπτυξη μια υγιού αγορά για startups κτλ. Παρ' όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει ένα στρατηγικό οικονομικό ανταγωνισμό. Αυτό θα μπορούσε να απορρεύσει από τι στρατηγικέ ε, επιχειρήσεων που θέλουν να κυριαρχήσουν στις διάφορε αγορέ ή όταν έχουμε ε, ηγετική θέση που αυξάνει την εθνική ισχύ. Αυτό αποτελεί πραγματικά μια μορφή κινδύνου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί αφορά ολόκληρα έθνη. Και αυτό μπορεί να ελεγχθεί υπό συμφωνίες Δηλαδή είναι μια στρατηγική βιομηχανική κούρσα τεχνητής νομοσύνης. Μετά έχουμε και τις ξεκάθαρες ε, στρατιωτικές ε, ανταγωνιστικές κούρσες για τα όπλα, για την ανάπτυξη ε, νέων οπλικών συστημάτων κτλ. Και αυτοί είναι ε, κίνδυνοι που θα μπορούσαν να α, ελεχτούν μέσω πούμε, συμφωνιών. Οι ανταγωνισμοί και οι κούρσες ανταγωνισμών για, ιδιαίτερα για τοπικά συστήματα θέτουν, σε μεγάλους, ε, θέτουν κίνδυνους διασπατάληση πόρων και θα μπορούσαν αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα αλλού. Στο ναυτικό, στα συμβατικά όπλα, στα πυρηνικά όπλα, ισχύει αυτό. Δεύτερον, ο φόβος για την απώλεια εθνικού πλεονεκτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει λοιπόν σε κάποιες πρακτικέ πρακτικές κλειδώματος διασφάλισης της ε, τεχνητής η οποία δεν θα μπορεί να ελέγχεται. Και τη στιγμή που είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία, όποιο ελέγχει την ε, τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καθορίσει πάρα πολλέ εξελίξεις ε, προ όφελός του. Οι ΕΠΑ φοβούνται θα χάσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα από την Κίνα. Και βέβαια αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, σημαντική ζημιά για τον υπόλοιπο πλανήτη. Επίσης θα μπορούσαν να έχουμε διαμάχες οι οποίες θα συνεχίζονται. Θα μπορούσε να υπάρχει μια αυτοτροφοδοτούμενη ε, ένα αυτοτροφωμένο κλίμα φόβου και δεν θα αναπτύξουμε την τεχνητή νομοσύνη για το κοινό καλό και αυτό ήδη το βλέπουμε να ισχύει από σήμερα. Τέταρτον και πιο σημαντικό ενδεχομένω, αυτέ οι δυναμικέ θα μπορούσαν να εκθέσουν τον κόσμο σε καταστροφικέ δράσει, επειδή ακριβώ θα αρχίσουν οι διάφοροι ισχυροί παράγοντε να περιορίζουν στον τομέα της ασφάλειας και να επηρεάζει αυτό την μακροχρόνια ασφάλεια των συστημάτων. Φανταστείτε λοιπόν όπου στο μέλλον αυτόνομα απλικά συστήματα θα αμήνονται υπέρ των δικών μας συστημάτων. Παρ' αυτά, αν μια ταχαία απάντηση είναι απαραίτητη, τότε θα πρέπει να έχουμε αυτά τα αυτόνομα, αυτόνομης ανταπόκριση συστήματα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και πολύ γρηγορούς ε, πολέμους. Ίσως να σκεφτούμε ότι αυτός ο κίνδυνος είναι μάλλον απίθανο να συμβεί. Όμως, να θυμάστε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η ΙΠΑ και η Σοβική Ένωση δημιούργησαν συστήματα πυραυλικά που έφταναν μέχρι το διάστημα. Πέμπτο στοιχείο που θα ήθελα να θίξω. Γιατί αυτοί οι εξοπλισμοί και οι κούρσει των εξοπλισμών είναι επικίνδυνοι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι πέραν αυτών που ανέφερα. Δηλαδή η διάβρωση των αξιών μας επειδή ακριβώς ε, έχουμε ε, εμπόριο αυτών των συστημάτων. Μπορεί ας πούμε οι χώρες να δουν ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα μπορούσαν να εμπορευτούν προσωπικά δεδομένα υπέρ ας πούμε, της ασφαλείας τους. Αυτά είναι λοιπόν κάποιες από τις ανησυχίες. Τι κάνουμε τώρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Θα είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε από μόνα τους, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καταρχάς θα μπορούσαμε να έχουμε σωστούς κανόνες και νόμους σε επίπεδο στόχων. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μέσω κανόνων, πρωτοβουλειών, της διαφάνειας, της ισότητας, στα αυτόνομα οπλικά συστήματα κυρίως. Όμως αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει αβεβαιότητα για το χαρακτήρα αυτού του προβλήματος και για το τι προσπαθούμε να αποφύγουμε. Οι λύσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να επινοήσουμε μπορεί ενδεχομένω να μην αρκέσουν για να αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους κινδύνους που ανέφερα προηγουμένως. Θα πω και δύο λόγια, σύντομα, μετά από αυτό που είπαν οι προηγούμενοι εισηγητές για τα εξοπλιστικά συστήματα και την εξέλιξη τεχνολογίας. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα φαινόμενα τα οποία είναι δύσκολο να ελέγξουμε είναι αυτά ακριβώς που έχουν προβλήματα συμμόρφωσης όσον αφορά την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης γιατί υπάρχει δυσκολία το να, στο να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε γιατί είναι αμοιβαία ωφέλιμο. Εξάζεται γρήγορα και η τεχνολογία. Ε, έχουμε και συμφέροντα όχι μόνο στα ειδικά, αλλά βεβαίω οικονομικά εξωτερικά συμφέροντα. Όταν λοιπόν αλλάζουν όλα αυτά ταχύτατα και ε, εμπλέκεται η τεχνολογία, τότε είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Αυτές είναι λοιπόν οι δυσκολίες, οι οποίες είναι ορατές και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε και συγκεκριμένε λύσεις. Η τεχνική νομοσύνη παρέχει δυνατότητες και αυτό ταυτόχρονα μας παρέχει κάποιες λύσεις. Ας πούμε θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου πολύ μεγάλο κομμάτι από το hardware θα περιέχει ένα δικό του σύστημα επαλήθευσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και συγκεκριμένα, αλλά και με κάποια δόση φαντασία, φανταστείτε έναν κόσμο που θα έχουμε αυτόνομα οπλικά συστήματα, τα οποία θα συνοδεύονται με hardware, το οποίο θα ανταποκρίνεται μόνο σε συντεταγμένες άμυνα. Φανταστείτε λοιπόν μια κατάσταση όπου η μία χώρα δεν θα φοβίζει την άλλη, δεν θα αποτελεί φόβητρο ή πιθανή απειλή για την άλλη. Θα πρέπει να έχουμε συνολικές, ολιστικές λύσεις για αυτές τις απειλές. Μπορούμε, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό μέσω διοχέτευσης αυτού του ανταγωνισμού για τον εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντω αυτός ο ανταγωνισμός διαβρώνει τις αξίες μας. Μπορούμε όμως, μπορούμε όμως ένα κομμάτι των πόρων μας να το διοχετεύσουμε υποστηρίζοντας αυτούς τους φορείς που προσπαθούν να ζητήσουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Οι πόροι μας, ας πούμε, οι οποίοι είναι ε, κοινοφελείς, όπως ε, χρηματοδότηση ε, ερευνητών, ταλέντων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτές, αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν λοιπόν να στηρίξουν αυτούς τους φορείς οι οποίοι δρούν υπέρ του κοινού καλού εις βάρος αυτών που δεν το κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε και τι, τι σημαίνει το να δράσουμε υπέρ του, υπέρ του κοινού καλού, ώστε να, α, οι δράσεις μας να είναι επικεντρωμένες και να έχουν νόημα. Κάθε φοράς λοιπόν θα πρέπει, που εμπλέκεται, θα πρέπει να μας εξηγεί το πώς ακριβώς βλέπουν τον εαυτό τους και τι ποιο είναι το, κινητό, το κίνητρό του. Επειδή εδώ δεν θα πρέπει μόνο να θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά να εξηγούμε και για ποιο λόγο το κάνουμε. Και ως πρώτο βέμα, θεωρώ ότι, ως, ε, καταρχάς μάλλον θέλω να πω, ότι αυτοί που αποφελούνται περισσότερα από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοί που λέγουν περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι περισσότερο υπόλογοι. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τον την κούρσα των, το εξοπλισμών από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια μοναδική πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Κίνα ή τη ΣΥΠΑ. Γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν κανόνες και θεσμούς που περιέχουν και κοινωνικές αξίες. Βρίσκεται λοιπόν στον κατα... στο... στο καταλληλότερο στην καταλληλότερη θέση για να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντα το διεθνή διάλογο, κάτι το οποίο αποτελεί το κυριότερο ε, στοιχείο για την επιβολή ακριβώ ε, προγραμμάτων, ε, προτύπων και προδιαγραφών. Και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σημείο του αιώνα που διατρέχουμε θα είναι ακριβώ ο έλεγχο αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη, στο να αποφύγουμε τι κοινωνικέ ταραχέ και αρνητικέ επιπτώσει, Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση και άλλων παγκοσμίων θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα έχει η διακυβέρνηση τη τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό θα πρέπει να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο οι κυβερνήσει. Ευχαριστώ πολύ. Well deserved applause. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας που ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ ε, σημαντικά. Ο κύριος Δίκοφ τώρα που είναι υπεύθυνος ε, του Τμήματος Ασφαλείας από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα να πω ότι θα εκφράσω προσωπικές ε, απόψεις ε, ως ε, επικεφαλής του Ιδρύματος Επιστημών και Πολιτικής και αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις όσον αφορά το iPro, το οποίο δεν θα το εκπροσωπήσω σήμερα, ε, ευχαρίστω ε, να τις ακούσω κάποια άλλη στιγμή. Ε, μπορείτε να δείτε βέβαια τις εκθέσεις του iPro στο διαδίκτυο, στο iPro.org. Κάποια στοιχεία των εκθέσεων αυτών θα τα αναφέρνω αυτά τα αναφέρω. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την άμυνα και στις εφαρμογές στο μέλλον. Ε, η τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη ε, θα βοηθήσει την ενίσχυση αυτόνομων λειτουργιών όπως ε, η στόχευση, η επιλογή, η εμπλοκή, η επίθεση θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, στα ε, διάφορα ε, σώματα, στην επιμελητεία, στη διοίκηση και τον έλεγχο. Είναι σαφές ότι η τεχνολογία και η εφαρμογή θα ρυθμίζεται σε κάποιο βαθμό, από ε, το στερεωτικό τομέα, από τα κράτη, από τους οργανισμούς ε, πιστοποίησης, από συμμαχίες, ε, υπό, διεθνή, το, υπό τη διεθνή νομοθεσία, όπως έχει γίνει και ως τώρα. Ένας λόγος όμως για τους οποίους διαφέρει αυτό, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι η δυνατότητά τους να λάβουν αποφάσεις για το πώς, αν και πότε θα χρησιμοποιηθεί η ισχύς με αποτέλεσμα ζωή ή το θάνατο κάποιων ανθρώπων. Αυτό λοιπόν θέτει κάποια ε, ηθικά ζητήματα και ε, ε, αποτελεί, δημιουργεί κάποια όρια για την νομοθεσία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για τον τομέα των φωνικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων, που είναι η σκληρή τεχνολογία και θα μιλήσω και για τη σύμβαση για τα συμβατικά όπλα ε, η σύμβαση αυτή δεν είναι το μόνο διεθνές, ο μόνος διεθνής φορέας ε, που ε, συζητά την ομοθεσία, την, τα όπλα αυτά, τα φωνικά όπλα. Από τη μία λοιπόν υπάρχει το θέμα των φωνικών αυτών ομονοπλικών συστημάτων. Από την άλλη όμως η σύμβαση αυτή είναι το κέντρο βαρύτητας όταν πρόκειται για την αμική, την νομική αξιολόγηση ορισμένων ζητημάτων εν ολίγης. Αυτά πρέπει να γνωρίζουμε σε σχέση με συζητήσεις, διαδικασίες, ορολογίες και ε, νομικά στοιχεία στο πλαίσιο της σύμβασης. Υπάρχει μία ομάδα κυβερνητικών ελέγχων που διερευνά τις, τους πιθανούς ορισμούς. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει πρόοδος σε σχέση με την εντολή. Κατά πάσα πιθανότητα οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν τη συζήτηση το 2019. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό των φωνικών αυτών ομονοπλικών συστημάτων, ούτε υπάρχει συμφωνία κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα οπλικά συστήματα ή όχι. Κάποια βέβαια κράτη, όπως είπα και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν τέτοιους ορισμούς. Η Σύμβαση για τα Συμβατικά Όπλα είναι ένα φόρουμ διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, Επομένως, ασχολείται με την ε, νομικώς αποδεκτή χρήση των οπλικών συστημάτων και όχι με τη ρύθμιση της τεχνολογίας. Αυτή η προσέγγιση που βασίζεται στο διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο ξεκίνησε μια συζήτηση κατά πόσο χρειάζεται ο όρος φωνικός ε, στα φωνικά αυτόνομα οπλικά συστήματα. Έχει όμως ε, διατηρηθεί για λόγους ε, συνέχειας. Καλύτερα να μιλάμε για αυτόνομε λειτουργίες στα οπλικά συστήματα και όχι για αυτόνομα οπλικά συστήματα για να μην γίνεται ανθρωπομορφισμός ε, των ικανοτήτων των, μηχανικών, των, ε, μηχανών. Για παράδειγμα, το Apple χρησιμοποιεί το σύστημα υπολογιστικής, υπολογιστικά συστήματα, για να τονίσει τη σημασία των ε, υπολογιστικών τεχνικών, για να μην χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως το σύστημα αποφασίζει, σκέφτεται κλπ. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να εκχωρήσουν αποφάσεις και καθήκοντα σε μία μηχανή. Ε, επειδή είναι επίμαχη τεχνική ορισμή και όχι εφικτή, η Σύμβαση για τα Συμβατικά Όπλα βασίζεται στο ανθρώπινο στοιχείο, εστιάζεται στο ανθρώπινο στοιχείο, στον έλεγχο των οπλικών συστημάτων. Ο διοικητής ε, ε, ε, ε πρέπει να κάνει την απαραίτητη κρίση όταν πρέπει βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε σχέση με την χρήση ισχύω. Αυτές είναι οι κρίσιμες λειτουργίες ενός οπλικού συστήματος. Το θέμα είναι πώς πρέπει να προγραμματίσουμε να εφαρμόζεται ή να ασκείται ο ανθρώπινο έλεγχο επί των οπλικών συστημάτων ε, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ε, στο επίκεντρο αυτών, ε, αυτής της ε, συμμόρφωσης υπάρχει η διάκριση μεταξύ των μάχημων και των μη μάχημων, η στρατιωτική αναγκαιότητα και αναλογικότητα της χρήσης ισχύω, όπως επίσης και η πρόληψη πριν από την εμπλοκή. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η έννοια του ανθρώπινου ελέγχου εξελίσσεται σε, ένα επιπλέον, σε μια επιπλέον αρχή που βασίζεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στο μέλλον. Τώρα, Τώρα, ο αντίκτυπο τη τεχνολογία για τι επιλογέ. Όπω είπα, η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο για την ε, ρύθμιση, έμεσα ή άμεσα, σε αντίθεση με άλλε ρυθμίσει για τα οπλικά συστήματα. Μεταβλητέ όπω ε, το υλικό, οι ορισμοί που έχουν να κάνουν με το υλικό, αριθμό των όπλων, τα είδη των όπλων δεν είναι επαρκεί παράγοντε. Είναι εύκολο, για παράδειγμα, να ορίσει κανεί ένα λέιζερ, ε, να μετρήσει κανεί τα κύρια άρματα μάχη, της ε, ή να παρουσιάσει, να περιγράψει έναν από θαλάσσις ε, εκτοξευόμενο πύραυλο, όμω είναι πολύ δύσκολο να ταξινοποιήσει ένα πνικό σύστημα με λειτουργίες αυτόνομες, ε, γιατί υπάρχει ο κύκλος στόχευσης. Ο δυναμικός κύκλος στόχευσης του iProw έχει έξι βήματα και αυτά είναι τα πιο σημαντικά εντοπισμός, καθορισμός, ανείχνευση, στόχευση, εμπλοκή και αξιολόγηση του αντικτύπου. Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι οι υπολογιστικές μέθοδοι όπως η εκμάθηση των μηχανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τμήμα του κύκλου στόχευσης. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ε, που αποτελούν συστήματα, όχι πλατφόρμες οι ευφυείς ή εν πάση περιπτώσει οι προηγμένες λειτουργίες τους μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ίδιο το μέσο κρούσης αλλά ε, μπορεί να ε, υπάρχει και στο δίκτυο των αισθητήρων, των επεξεργαστών, των πλατφορμών κλπ. Ε, υπάρχουν ικανότητες που αναπτύσσονται με την πολλαπλότητα της δικτύωσης και όχι με μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Υπάρχουν οι ομάδες οι επανδρομένες ή μη επανδρομένες που προσθέτουν τον ανθρώπινο παράγοντα στην εξίσωση, αλλά ο ανθρώπινος ρόλος μπορεί να ποικίλει από παρακολούθηση μέχρι καθοδήγηση. Είναι εύκολο να πει κανείς ότι υπάρχει ένα επανδρομένο σύστημα ή ένα τηλεκατευθυνόμενο σύστημα, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε ένα πλικό σύστημα με αυτόνομες λειτουργίες, ε, γιατί υπάρχει και λογισμικό. Και όταν γίνεται η δοκιμαστική χρήση αξιολόγηση των, αξιολόγηση των εκατοτήτων αυτών, τα δεδομένα και το ε, πλαίσιο είναι σημαντικά, όπως ο κώδικας, για παράδειγμα, και η, ε, ισχύς επεξεργασίας. με την εκμάθηση της μηχανής, η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων είναι αυτό που αλλάζει την κατάσταση. Υπάρχει μια ηθική και δεοντολογική ε, πτυχή ε, το να Όσο ε, ε, προς την ηθική διάσταση υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες που συζητούνται στη σύμβαση για τα συμβατικά όπλα. Υπάρχει το επιχειρησιακό κομμάτι, είναι η σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή ε, υπάρχει μια έκθεση σχετικά του Μαρτίου του 2018. Σε πραγματικό επίπεδο ε, είναι ένα ισχυρό κίνητρο να μην υπάρχει ε, να μην υπάρχουν απώλειες από φίλια πειρά στις στρατιωτικές στην στρατιωτική ισχύ και για το προσωπικό και για τον εξοπλισμό. Αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση και με την ακρίβεια του στόχου και με την πρόληψη και με την ε, αποτελεσματικότητα. Ε, ο στρατιωτικός τομέας χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς για να επιτύχει τον έλεγχο της ε, βίας ε, τα προηγμένα όπλα έχουν διάφορες, ε, διάφορους τρόπους λειτουργίας, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ασφαλείας, υπάρχει εκτεταμένο ε, σχεδιασμός που εξασφαλίζει τον τρόπο με τον οποίο δεν έχουμε απώλειες από φίλια πυρά και βέβαια στο πλαίσιο κάποιων νομικών προδιαγραφών για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι είναι στρατιωτικό πλεονέκτημα να υπάρχει έλεγχος επί της χρήσης ε, των ε, δικών μας οπλικών συστημάτων πρέπει να είναι ε, προβλέψιμα και αξιόπιστα για να υπάρχει ε, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει και το νομικό κομμάτι. Το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο είναι η νομική βάση στις συγκρούσεις. Παρόλα αυτά ε, δεν έχουν πλήρως αποσαφινιστεί τα κάποια στοιχεία, όπως το επιπρόσθετο πρωτόκολλο στην Σύμβαση της Γενέβη. Χρειάζεται πάντως μία ανθρώπινη κρίση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση βίας για τεχνικούς και νομικούς ε, λόγους δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθεί αυτό στις μηχανές. Επίσης, η σωστή ανθρώπινη κρίση σημαίνει ότι καταλαβαίνει καλής καλά μια κατάσταση και αυτό αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης. Μόνο η εμπλοκή των ανθρώπων στην διαδικασία στόχευσης και την ικανότητα ε, του διοικητή να παρέμβει κατά τη διάρκεια ε, των ε, επιχειρήσεων ε, εξασφαλίζει την ευθύνη και τη λογοδοσία στο πλαίσιο της στρατηγικής ιεραρχίας. Τρίτο στοιχείο, διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Ήδη σήμερα η τεχνολογία έχει επιτύχει αυτόνομες λειτουργίες στα οπλικά συστήματα και υπάρχει συνεχής διάδοση. Ένας από τους λόγους είναι η επιστήμη, η βιομηχανία, τα κράτη κάτι το οποίο όλοι ε, λέμε ότι το υποστηρίζουμε και δεν θέλουμε να το ρυθμίσουμε, αυτό καθεαυτό. Όμως ε, η ενίσχυση των στρατιωτικών πλεονεκτημάτων όπως μια καλύτερη ακρίβεια και μια μεγαλύτερη ταχύτητα επίθεσης και μάχης είναι επίσης σημαντικά. Συνεπώς υπάρχουν ε, προγράμματα στρατηγικής ανάπτυξης και προγράμματα ε, εξοπλισμού ε, για τα αυτόνομα συστήματα και την τηλεκατεύθυνση. Αυτό υπάρχει, ασχετίζεται με μία τάση στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέμε ότι είναι η δυναμική των εξοπλισμών, για παράδειγμα στα κράτη P5, που ε, παράλληλα έχουν κάποιους συνδυασμού ω προς την ρυθμιστική προσέγγιση της ε, σύμβασης ε, για τα συμβατικά όπλα. φοβούνται την κλιμάκωση της κρίσης και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση, των κρίσεων και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Θα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της ε, ταχύτητας στο πεδίο μάχης που θα συνδέεται με, ένα, μια, μια απώλεια επιχειρησιακού ελέγχου. Υπάρχει και το ηθικό ε, ζήτημα. Είναι δυνατόν να, να εκχωρήσουμε σε μια μηχανή το, την, την απόφαση για ζητήματα ζωής και θανάτου. Ε, σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα ζήτημα ε, στην άμυνα έχει να κάνει με την ε, ηθική θεωρία που ισχύει. Η τελευταία έκθεση του IPRAU θεωρεί ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ο βασικός παράγοντας. Ε, δύο ε, ζητήματα υπάρχουν για τη διερεύνηση των συνεπειών μιας ενδεχόμενης ρύθμισης. Η αυτονομία των οπλικών συστημάτων ε, διασπά τη σχέση με την ηθική και πράγματι παραβιάζει την ε, αξιοπρέπεια του θύματος και μπορεί οι συνέπειες, δηλαδή το αναμενόμενο πλεονέκτημα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ε, ή χρήσης ισχύω στο συνδυασμό με, τα με τις αυτόνομες λειτουργίες να ε, παραβιάζουν ζητήματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το iPro καταλήγει στο εξή αποτέλεσμα. Ανάλογα με την ηθική μας θέση θα ε, έλεγε κανείς ότι μπορεί να μην υπάρχει αυτή η σχέση ε, με την ηθική λόγω των αυτόνομων λειτουργιών, ότι δηλαδή καλό θα ήταν να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ηθική, θα μπορούσαμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε τη χρήση του οπλικού συστήματος το πλαίσιο μιας ηθικής, κάτι το οποίο θα σήμαινε ανθρώπινος έλεγχος και στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό αλλά και στη χρήση. Υπάρχει δηλαδή αναγνώριση, σιωπηρή ή σαφής, της αρχής του ανθρώπινου ελέγχου. Να σας πω τώρα το συμπέρασμά μου. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν σημαντικά κίνητρα και... Ε, λόγοι ρύθμισης των ε, φωνικών αυτών οπλικών συστημάτων μπορεί να μην γίνεται λόγω του ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ορισμοί το συζητάει η Σύμβαση για τα, για τα συμβατικά όπλα, για τη ρύθμιση της χρήσης αυτών των όπλων. Ε, μεγαλύτερη ρύθμιση θα σήμαινε επίσης ε, και ότι αυτό θα διέπει και το σχεδιασμό και τη δοκιμή ε, των συγκεκριμένων συστημάτων, ε, ζητούμε δηλαδή στο επίπεδο του ΆΙΠΡΑΟ μια θετική ρύθμιση με ανθρώπινο έλεγχο ε, στο σχεδιασμό και τη χρήση των οπλικών συστημάτων, δύο κριτήρια για την διασφάλιση του ανθρωπίνου ελέγχου, έλεγχος ε, μέσω του ελέγχου και κατά τη χρήση και από την άλλη κατανόηση της κατάστασης και δυνατότητα παρέμβασης για τον διοικητή ή τον χρήστη ενός συστήματος από την άλλη η αναθεώρηση των όπλων ε, που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 36 του επιπρόσθετου πρωτοκόλου της Σύμβασης της Γενέβης λέει ότι η αξιολόγηση και η δοκιμή των όπλων είναι κάτι απαραίτητο, αλλά δεν είναι επαρκές για τη διατήρηση του ελέγχου, του ανθρώπινου ελέγχου. Χρειάζεται και μια, ένα πλαίσιο ηθικό δεν πρέπει ο ανθρώπινος έλεγχος να αντικατασταθεί από την εισαγωγή τέτοιου είδους λειτουργιών στις μηχανές και στα συστήματα. Δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινου ελέγχου όσον αφορά τη χρήση ε, στην επιμελητία, τη μυστικέ υπηρεσίε, τι μυστικέ πληροφορίε και σε άλλου τομεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, όμω ε, ένα απαραίτητο όρο για την υπεύθυνη χρήση όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία σε σχέση με τους αλγόριθμους υπάρχουν ακόμη και στις αυτόνομες λειτουργίες των οπλικών συστημάτων ε, που μπορεί να ενισχύσουν την ακρίβεια σε ε, πολύ αυτοματοποιημένα μεντικά συστήματα μπορεί να γίνει αυτό. Υπολογιστικές μέθοδοι μπορεί να ε, αμφισβητήσουν τον ανθρώπινο έλεγχο στα οπτικά συστήματα. Ο σχεδιασμός και οι επιχειρησιακές διαδικασίες όπως και η κατάρτιση του προσωπικού πρέπει να εξισορροπεί και να περιορίζει αυτές τις τεχνικές ε, σε ένα βαθμό που είναι σε πραγματικό χρόνο κατανοητός για τους ανθρώπους, ε, τους χειριστές και τους ε, διοικητές. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρχεται τώρα η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη, τα πολύ ακριβή στοιχεία που μας έδωσε σε σχέση με την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Δυστυχώς είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση και απουσίαζα στην αρχή. Πριν από 10, χρο... πριν από 10 μέρες ήρθα σε επαφή με γερμανούς διπλωμάτες ε, και μας είπαν ότι υπάρχουν διεθνείς διαπραγματεύσεις για τα αυτόνομα ε, συστήματα, αλλά υπάρχει και ένα think tank, το SWP στη Γερμανία, που ασχολείται με αυτό το θέμα, ε, με τα ζητήματα που πραγματεύεστε κι εσείς. Είναι σημαντικό που έχει δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια όχι ακόμη. Αυτό είναι ενδιαφέρον, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, κυρία Άντερσεν στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μία από τις χώρες που δεν ήθελε να υπάρξει ένα πλαίσιο διεθνούς νομοθεσίας είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. και Υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε σε κάποιο είδους νομική συμφωνία ότι αυτά τα οπλικά συστήματα πρέπει για παράδειγμα να ε, απορριφθούν γιατί για μας είναι ένα ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει έρευνα ε, και ανάπτυξη, 13 δις ε, από το 2021 στο 2027 θα διατεθούν και εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να είναι σαφές ότι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα δεν θα ε, συμπεριληφθούν παρά ε, το ε, γεγονός ότι κάποιοι είναι υπέρ σε μεγάλο βαθμό. Είναι διαφορετικές, είναι διαφορετικές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετικά βλέπουν τα πράγματα. Εσείς πώς βλέπετε την Αμερική στη συζήτηση αυτή στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλε χώρε η Κίνα, η Ρωσία που αναφέρθηκαν σήμερα και επίση ενδιαφέρονται για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πώς καλύπτουμε λοιπόν αυτό το ε, ε, χάσμα. Όχι αυτόνομα οπλικά συστήματα, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που με ε, τρόπο που να μπορούμε να έχουμε ένα έλεγχο σε αυτήν την κούρσα. Νομίζω ο συνάδελφος θα πρέπει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσω και την ερώτηση του κυρίου Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους μας. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, στο παρελθόν, κατά τον ψυχρό πόλεμο, ο περιορισμός της κουρσα των εξοπλισμών ήταν ε, δυνατός μόνο και, όταν και οι δύο πλευρές καταλάβαιναν ότι το να μην κάνουν κάτι θα είναι ε, κακό για τους ίδιους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση ή τέλος πάντων την ανάλυση, ποια είναι η ανάλυση σας σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία. τι θεωρείτε ότι είναι ένα πιθανό σημείο αφετηρίας για μια αρχική συνεννόηση, γιατί αν μια πλευρά θέλει να προχωρήσει, ε, τότε δεν μπορεί πρόκειται να γίνει τίποτα. Η δεύτερη ερώτηση. Είχαμε μία συζήτηση για αυτά τα φωνικά αυτόνομα απλικά συστήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αντιπρόεδρος ε, και πατή εκπρόσωπος ε, Φεντερίκα Μογκερίνη μας είπε κάποια πράγματα αλλά δεν ε, είναι, μια, δεν είναι τεχνική εμπειρογνώμονας που να έχει μια σημαντική θέση ως προς αυτό. Εσείς πώς βλέπετε ότι είναι η κατάσταση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωση ώστε να υπάρχει ο απαραίτητο δημόσιος διάλογος. Και τρίτη ερώτηση. Υπάρχει κάποιο όριο για το οποίο θα λέγατε ότι είναι μια κόκκινη γραμμή, ότι εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Παρουσιάσατε και οι δύο διαφορετικές στρατηγικές ε, και ε, διαφορετικές συζητήσεις, όμως Υπάρχει κάποιο όριο που να πρέπει να τεθεί σε αυτήν την ε, εξέλιξη ώστε να μην μας ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου και θα μπορούσε αυτό το σημείο να είναι η βάση για πρόοδο και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να ε, εκμεταλλευτώ τη θέση μου ως Προεδρού και να παρέμβω, όμως ε, πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ε, δίλημα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε όλοι σας όσον αφορά τις διάφορες εντάσεις που υπάρχουν σχετικά με αυτή την κούρσα το να είσαι ο πρώτος, ο καλύτερος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την ιδέα ότι περιμένουμε, δημιουργούμε συστήματα ασφαλείας, νομοθετούμε. Όμως αναφερθήκατε επίσης όλοι σας, και αυτό σχετίζεται με την τελευταία ερώτηση, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης λόγω της ε, φήμης μας, του πώς μας βλέπει ο κόσμος. Και σε αυτό το πλαίσιο και επειδή μιλάμε για τις εξερίξεις στον πυρηνικό τομέα, ίσως το σημείο καμπής να ήταν η κρίση στην Κούβα και ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα ατυχήματα, αυτές τις εντάσεις Και σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρομαι πολύ για την πρότασή σας κύριε Νταφά ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σώμα που θα αξιολογεί, θα φέρνει σε επαφή τους ε, ράγοντες, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα μπορούσατε ίσως να γίνετε πιο αναλυτικός πάνω σε αυτό. και θα μπορούσε όλο αυτό ίσως ε, κατά τη γνώμη σας να ενσωματωθεί και σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Ε, αυτό το οποίο δεν κάνω είναι να μιλάω κάτι για το οποίο δεν ε, γνωρίζω πολλά και γι' αυτό το λόγο θα δώσω το λίγο στον κύριο Νταφό. δεν θέλω να φανταστώ κάτι, να δημιουργήσω κάτι απλά και μόνο για να φανώ έξυπνη. τότε ε, θα στραφώ πρώτα προς τον ε, κύριο Τίκο ε, και στη συνέχεια κύριε άμα μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, υπάρχουν ορισμένα Εθνικά Κοινοβούλια τα οποία έχουν λάβει αποφάσεις πάνω στο θέμα, όπως για παράδειγμα των κάτω χωρών, Δεν γνωρίζω τι αποφάσει και αν υπάρχουν σε Γαλλία και Γερμανία. Υπάρχουν συζητήσει μεταξύ των βουλών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ε, έγινε, ε, όπου έγινε έτοιμα να υπάρξει ένας νέος ορισμός σχετικά με το τι είναι τα όπλα αυτά. η κυβέρνηση κάνει μια συζήτηση λοιπόν. Υπάρχει παρόλα αυτά μεγάλη, μεγάλος δρόμος μπροστά μας γνωρίζω ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ε, για αυτή την ε, συζήτηση ε, σε επίπεδο επιτροπής όπως εδώ η έτσι και στη Γερμανία γίνονται ακροάσεις αλλά βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Μπουτικόβα που είναι το κοινό έδαφος για νομοθεσία. τουλάχιστον όσον αφορά τις συζητήσεις του CCW επαναλαμβάνουμε και δίνουμε έμφαση ε, στο ε, να υπάρχει ανθρώπινος όλων, έλεγχος των, των οπλικών συστημάτων και αυτό αφορά ειδικά τα επίπεδα όπου υπάρχει δισταγμός ε, εισαγωγής νέων ε, νομοθετικών εργαλείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είναι ε, η πρώτη που το τονίζει αυτό πάντοτε έχουν έλεγχο των οπλικών συστημάτων Ορισμένες χώρες ίσως θα δίσταζαν να συμφωνήσουν ότι ήδη υπάρχει μια αρχή ανθρώπινου ελέγχου, τουλάχιστον σε αναπτυξιακό στάδιο. Όλοι αναφέρονται σε αυτό το στάδιο ως εθνική κατευθυντήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι το κοινό έδαφος είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει να χάσουμε τον έλεγχο των οπλικών μας συστημάτων όπως η κρίση ε, της ε, Κούβας είναι όταν, ε, όταν θα έχουμε δύο συστήματα τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε το ένα οπλικό σύστημα με το οπλικό σύστημα ενός μιας άλλης χώρας. Αυτός, αυτή είναι η φύση του πολέμου. Οπότε βρισκόμαστε ε, σε μια κατάσταση όπου κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο. διότι η μάχη σε ταχύτητα μηχανής γίνεται έτσι που δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει καν τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή, κατά τη γνώμη μου λίγο πιο πριν, Αυτά λοιπόν είναι ένα από τα σενάρια όπου ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν ε, σοβαροί κίνδυνοι. Τώρα όσον αφορά το ρόλο της ε, Ρωσίας και της Κίνας, είναι δύσκολο να καταλάβουμε την Ρωσία. Η Κίνα εξέπληξε την ε, διεθνή κοινότητα πέρσι με μια πρόταση νομοθέτησης ε, και απαγόρευσης αυτόνομων μονοπλικών συστημάτων και ακόμα πρότεινε και ε, κριτήρια σχετικά με το τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα. Όμως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν αυτά θα πρέπει να ισχύουν όλα τα κριτήρια ή μονάχα ένα από τα πέντε και αυτό το οποίο πρότειναν είναι μια απαγόρευση της χρήσης αυτών των συστημάτων, οπότε με βάση αυτό ο καθένας θα μπορεί να τα αναπτύξει, αλλά όχι να τα χρησιμοποιήσει. Δεν υπήρξε επίσημη ανταπόκριση από άλλες χώρες ε, πάνω σε αυτή την πρόταση. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά ε, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα φόρα, όμως ε, μέχρι στιγμής δεν έχει μια κοινή θέση. Και τέλος, όσον αφορά το τελικό ερώτημα, σχετικά με το πώς θα ρυθμίσουμε την ε, πολιτική διαδικασία εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, για το οποίο όμως δεν έχω μια καλή απάντηση. Η απόφαση του Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα βοήθησε διότι ε, συνέβαλε σε μια ευρύτερη συζήτηση ε, όσον αφορά τις ηθικές προκλήσεις ε, όσον αφορά αυτή την τεχνολογία γνωρίζω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία διστάζουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα διότι δεν υπάρχει μια κοινή θέση των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη έχουν και διαφορετικά συμφέροντα. Όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ανταλλαγή ε, των, ε, μεταξύ των κρατών μελών ε, σε κοινό επίπεδο. Σίγουρα θα είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτό. Όμως το να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή θέση θα είναι δύσκολο. Όμως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα ήταν μια ε, για τα ε, υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες χώρες ε, να προσαρμόσουν αντιστοίχως τις ε, θέσεις τους ε, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε ομαλά και στον κύριο ε, Νταφό, ο οποίος ε, θα ε, μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα ήταν ωραίο αν είχα το σχεδιάγραμμα της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα. Υπήρξαν ενδιαφέροντα ερωτήματα και αποτελούν κίνητρο για να ζητήσουμε λεπτομέρειες και να το προωθήσουμε όλο αυτό. Και φυσικά ε, το ερώτημα είναι και το επίπεδο στο σε ποια φόρα θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβούλιο. Θα έλεγα μια γενικά ότι είναι πολύ νωρί όσον αφορά την διακυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή την οποία δεν θα πρέπει να περάσουμε μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένες νομοθεσίες ε, όσον αφορά τους στόχους, ε, ποιες θα είναι οι πολιτικές τις οποίες δεν κάνει να περάσουμε, για παράδειγμα. Ε, μπορούμε να προσπαθήσουμε και πρέπει. Όμως, εάν πιέσουμε πολύ για την τελική λύση, μπορεί να έχουμε το λάθος αποτέλεσμα να περάσουν ε, πέντε χρόνια και να αποτύχει η πολιτική αυτή. Α κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω και α επικεντρωθούμε καλύτερα ίσως ε, σε ε, λύσεις, μεταλύσει υψηλότερου επίπεδου. Θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, πολύ πιο σοβαρή συζήτηση από σήμερα, Αυτές οι συζητήσεις στα κοινοβούλια θα πρέπει να γίνονται καθημερινά ε, όπως ισχύει και με τη διακυβέρνηση ε, των πυρηνικών ε, όπλων το 45 και το 46 ήταν το βασικότερο θέμα το οποίο συζητούσε ο κόσμος πώς θα είναι ο πλανήτης πώς, όταν βλέπαμε τι θα γίνει με την Ευρώπη τότε το ζήτημα των πυρηνικών όπλων βρισκόταν στο επίκεντρο θα πρέπει να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο τόσο μεγάλο είναι το, το θέμα αυτό όμως, εάν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο από φόβο και πανικό, ε, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Για να έχουμε αποτελεσματική πολιτική θα πρέπει να έχουμε ε, λογικοί τεχνοκράτες οι οποίοι θα σχεδιάσουν ε, μια βιώσιμη πολιτική δεν μπορούμε να έχουμε ε, μια απλουστευμένη προσέγγιση και να λέμε ότι αυτό είναι κακό και η πολιτική χτίζεται γύρω από αυτό το κακό. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ε, δεν ε, θα πρέπει να έχουμε μια κατάσταση όπου ε, ο πληθυσμός φοβάται. Το βλέπουμε αυτό ήδη. Υπάρχει ήδη φόβος όσον αφορά τα εργασιακά και το πώς θα επηρεαστούν. Όμως θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο πληθυσμός και να είναι μια, μια πολιτική δύναμη την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε η οποία όμως ταυτόχρονα μπορεί να και ξεφύγει και εκτός ελέγχου και δεν θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια αποτελεσματική συζήτηση. Τώρα αν υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και πού μπορούμε να την ε, τραβήξουμε. Η αυτονομία στα οπλικά συστήματα μπορούμε να, εκεί να εξετάσουμε ποια είναι τα επικίνδυνα στοιχεία τα οποία πρέπει να σταματήσουμε. Η γενική μου απάντηση είναι ότι θα είναι δύσκολο. Οι εξελίξεις ε, στην ε, τεχνητή νοημοσύνη ε, είναι απότομες και δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε ε, κόκκινε γραμμέ. Ε, για παράδειγμα, τα γενικά συστήματα ή τα συστήματα τα οποία προσαρμόζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά καλύτερα ή όπω οι άνθρωποι. Ε, αυτό ίσω φαίνεται τρομακτικό. Ή συστήματα τα οποία ε, ενώνονται σε διάφορες, σε με διάφορα συστήματα. ίσως ε, θα θέλουμε να περιορίσουμε την νοημοσύνη ε, του συστήματος, να μην είναι πολύ νοήμων σε ορισμένους ε, τομείς ή σε επίπεδο που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να το καταλάβει. Αυτές όλες είναι διαστάσεις τις οποίες ίσως θα θελήσουμε να ελέγξουμε κατά την εξέλιξη όμως. Αν έχουμε καλά ε, διακυβερνητικά συστήματα δεν υπάρχει λόγος να το μπλοκάρουμε διότι είναι δυτή η χρήση. Μπορεί να οδηγήσει σε ε, βελτιώσει στον τομέα υγεία στην οικονομία. τέλος πώς θα είναι αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο προστατεύει τις αξίες μας. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει την επιτυχία αυτής της ε, πρωτοβουλίας είναι αν υπάρχει ε, τεχνική ηγεσία, ακόμα και στο πλαίσιο της διακυβέρνησης, ε, βοηθά αν υπάρχουν ειδικοί εμπειρογνώμονες πραγματικά ταλέντα, κάτι το οποίο έχει η Ευρώπη. Πολλοί δεν θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη, θέλουν να παραμείνουν, οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα εγχώρια συστήματα. Ε, ο κύριος Μακρόν το κατάλαβε αυτό καλά. Είναι το ζήτημα της εμπιστοσύνης ε, στο να είσαι μια ε, ηγετική δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Εάν για παράδειγμα η εμπιστοσύνη στο Facebook πέσει, αυτό επηρεάζει το επιχειρηματικό μοντέλο του Facebook. Καθώς επίσης ε, και το Facebook ως ε, έναν ηγέτη της, τεχνητική, της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε ε, θα πρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αυτό θα ήταν ένα ωφέλιμο στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο σωστός θεσμός, μπορεί να δημιουργήσει ε, κανόνες και να αποκτήσει μια φήμη ότι το κάνει αυτό για το κοινό καλό. Μπορεί να ξεκινήσει από μικρότερα προγράμματα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πιο πολύπλοκα Μπορεί να το κάνει αυτό για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άμα κοιτάει μακροπρόθεσμα και θέλει να γίνει το επίκεντρο παγκόσμια συνεργασία προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να το κάνει αυτό λαμβάνοντα υπόψη τη τα παγκόσμια συμφέροντα. Μπορεί να πει ότι το κάνει αυτό για το παγκόσμιο κοινό καλό. Και τα πλεονέκτημα και τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα έχει μια αξιόπιστη διάβγεια, διαφάνεια, ε, και ότι πραγματικά στοχεύει ε, για το κοινό καλό και ταυτόχρονα θα υπάρχει και διαφάνεια για τη δημιουργία ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή λοιπόν είναι η εξειδικευμένη αγορά στην οποία μπορεί να στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να είναι ένα ε, δημοκρατικός, ε, ένας δημοκρατικός διαφανής θεσμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να δημιουργήσει έτσι ένα καλύτερο σύστημα ε, τεχνητής νοημοσύνης που να χαίρει εμπιστοσύνη, όπως, όπως έχουμε το Fair Trade για παράδειγμα. Αν λοιπόν όλα αυτά πάνε καλά. Αυτό δεν είναι μονάχα καλό, αλλά μπορεί να αυξήσει τα πρότυπα ε, και για την Κίνα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για άλλα κέντρα ε, τεχνητή νοημοσύνη, ούτω ώστε να ανταγωνίζονται όχι μονάχα στην αποδοτικότητα και στην ε, δύναμη, αλλά ταυτόχρονα και στη διαφάνεια. Αν έχουμε αυτό το, αυτή τη δεξαμενή ε, δυνατοτήτων για την, καλή, για την καλή διακυβέρνηση, τότε μπορεί να γίνει ένα ανταγωνισμό για τα καλύτερα αποτελέσματα. Είχαμε αναφορέ στην πυρηνική τεχνολογία μετά το 45 και το 46 όταν ε, γινόταν σοβαρές συζήτησεις, ε, σοβαρές συζητήσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλικών συστημάτων ε, ίσως να το ξεχνάμε αλλά είχαμε εκείνη την στιγμή μόλις είχαμε βγει από έναν τρομακτικό πόλεμο και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δημιουργήσαμε τον ΟΗΕ. Ο Ρούσβελτ πραγματικά ήθελε να δημιουργήσει αυτή την παγκόσμια ειρηνική τάξη. Φτάσαμε κατά το ίμιση εκεί. Τα πυρηνικά όπλα αναγνώρισαν ήδη από τότε ότι η κούρσα των εξοπλισμών θα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θα ήταν αφελές να μην το πιστεύουμε αυτό. Όμως υπήρχε πίεση, πίεση ε, από επιστήμονες, από τους απλούς πολίτες. αλλά και από ιδεαλιστικές πολιτικές ελίτ που έλεγε ότι ε, εδώ είναι η ευκαιρία. Μια κούρσα θα είναι καταστροφική και έχουμε τη δυνατότητα να την ε, σταματήσουμε. Βρετανία, Σοβιετική Ένωση, είπα, ήταν ακόμα σύμμαχοι σε εκείνη τη φάση και σκέφτηκαν ωραία πώς θα το κάνουμε. Προχώρησε πολύ η συζήτηση, υπήρξε συζήτηση στον ΟΗΕ. Υπήρξαν διάφορες προτάσεις, το σχέδιο Brook ήταν ίσως κοινικό, όμως ε, υπήρξαν διάφορες αναφορές ε, και εκθέσεις που κάνανε καλές ε, προτάσεις όπου οι ΗΠΑ θέλαν, για παράδειγμα, να προστατεύσουν τα συμφέροντά του, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και παγκόσμιο έλεγχο των πυρηνικών ε, όπλων. Έτσι, βλέπαμε τι ΗΠΑ διατεθειμένε να εγκαταλείψουν το μονοπόλιο του όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Δεν είχε αποτέλεσμα και υπήρχαν διάφορες, διάφοροι λόγοι, όμω, ε, υπό άλλε συνθήκε θα μπορούσε να είχε επιτυχεί. Μπορούμε να λάβουμε μαθήματα από εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι δύσκολη να ελεγχθεί ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός ε, συγκρούονταν, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, οπότε ο έλεγχος δεν θα επιτύχαινε. Όμως σήμερα δεν έχουμε αυτό το επίπεδο εχθρότητας ε, ε, που είχαμε τότε. Υπάρχει μεγαλύτερη συμβατότητα σε οικονομικά συστήματα, σε πολιτισμούς και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε προχωρήσει στο να έχουμε ένα παγκόσμιο ε, πολιτισμό, υπάρχει κοσμοπολιτισμός, το οποίο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η πρόκληση που θα έχουμε είναι ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα επικίνδυνα κομμάτια από τα ειρηνικά οικονομικά κομμάτια. Θα πρέπει λοιπόν να ταυτοποιήσουμε το στομίσο που θα μπορούμε να έχουμε μονοπόλια Και βέβαια μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και μονοπερό τα ωφέλη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τόσο πολλά χαρακτηριστικά όσο η πυρηνική τεχνολογία. Όμως, παρόλα αυτά, ότι γεωπολιτικά και πολιτισμικά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες με την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν λοιπόν δημιουργήσουμε μία ε, αλυσίδα εφοδιασμού ε, υπάρχουν προκλήσεις, όμως μπορούμε να προσπαθήσουμε και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και αυτό θα μπορούσε να ήταν η βάση ε, του παγκοσμι... ενός παγκοσμίου ελέγχου, ακόμα και αν αποτύχει, όμως θα μπορούσε να είναι ε, μια βάση για την μη προώθηση τέτοιων συστημάτων. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις όμως κατά τη γνώμη μου η ιστορία του αιώνας μας θα είναι εάν ε, μπορέσαμε να ε, είμαστε επιτυχημένοι ε, σε αυτήν την πολιτική πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Και ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις ε, ομιλίες σας, ε, για τις απαντήσεις ε, που δώσατε. και ακούσαμε τις συστάσεις σας ώστε το θέμα αυτό να έρθει πιο πολύ στο επίκεντρο. Πιστεύω ότι και σήμερα σε σύγκριση με το 45-46 υπάρχουν προκλήσεις, όπως και να έχει. Πιστεύω ότι ε, βοήθησαν ε, ιδιαίτερα οι απαντήσεις και τα σχόλια ε, που κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ και θα ανταποκριθούμε των υποχρεώσεων μας.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 Right. <laughs> And this is the uh, Ωραία. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Με ένα πρώτο ενδιαφέρον τμήμα σήμερα το πρωί και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Μελλοντικές προκλήσεις για το Ευρωπαϊκό Κέντρο το δορυφορικό της Ένωσης. Έχουμε τον κύριο Πασκάλ Αγγέν και τον κύριο Νίκολο Στάσιν. Άρμο για θέματα πολιτικής στη μονάδα ψυχής ομάδας για το διάστημα διεύθυνση πολιτικής ασφάλειας. Καλώς ορίσατε και δυο σας. επειδή ακριβώ το ΙΟΥΣΑΤΣΕΝ υποστηρίζει την πολιτική άμυνα και ασφάλεια τη Ένωση, πολύ σημαντικό κομμάτι των πολιτικών τη Ένωση. Παρέχεται σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, δεδομένα σε σχέση, κρίσιμα δεδομένα για την ασφάλεια και την άμυνα και μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε σημαντικές, σημαντικά μέτρα ανθρωπιστικά και διπλωματικά έγκαιρα ώστε να σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις μας. Κύριε Λεγκέ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Πέρσι τον Ιούνιο είχατε έρθει. Εν μεταξύ, τα στήματα άγιες προειδοποίησης και τα δορυφορικά έχουν όλο και πιο μεγάλη αξία και σημασία για την ασφάλεια και την άμυνα, οπότε προσβλέπουμε να ακούσουμε από εσά δύο λόγια για το κέντρο βέβαια, τις υπηρεσίε του, τις δάσεις του, τη δουλειά σας στο παρελθόν και τώρα και τι προσδοκάτε, τι αναμένετε τους επόμενους 12-18 μήνες και συγκεκριμένα πώς εντάσσεται το EU SATSEN στην γενικότερη πολιτική, στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι αναμένουμε τη συμβολή σας και να ξέρετε επίσης ότι μεταδίδεται ζωντανά μέσω ίντερνετ η συνεδρίασή μας. Έχετε το λόγο κύριε Λέγκε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτά τα γενικά λόγια, τα προκατακτικά. Και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την υπηρεσία μας, η ΣΑΤΣΕΝ. Όπως είπατε, θα μιλήσουμε για τις μελλοντικέ προκλήσεις για το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την τωρινή κατάσταση πριν περάσουμε στο μέλλον. Το κέντρο μας λοιπόν στηρίζει την ε, Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας στις διάφορες δραστηριότητες πολιτικής της και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι ακριβώς είναι το δορυφορικό κέντρο, πώς διοικείται και πώς λειτουργεί. Η αποστολή του αποφασίστηκε από τις χώρες μέλη για να στηρίξει τις πολιτικές ένωσης στο τομέα άμυνας και ασφάλειας μέσω διαφόρων επιχειρήσεων και αποστολών παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες με την χρήση διαστημικών μέσων, κυριότερα δορυφορικών δεδομένων μέσω διαφόρων πηγών για να κάνουμε ακριβώς και να πέρα στην αποστολή μας. Οι δραστηριότητε μας είναι συνεχόμενες σε καθημερινή βάση όλο το 24ωρο σε διάφορα μέρη του κόσμου και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε κάποια αυτονομία δορυφορική. Έχουμε δύο επίπεδα διακυβέρνησης, διοίκησης. Ένα πολιτικό επίπεδο με πολιτική καθοδήγηση. Έχουμε την Επιτροπή Ασφάλειας που μας παρέχει τους κυριότερους προσανατολισμούς και κατευθυντές γραμμές και έχουμε ένα λειτουργικό επίπεδο, επιχειρηματικό επίπεδο. Η κυρία Μογκερίνη αποτελέσουμε την ηθήνουσα αρχή μας εδώ. Και ο, λο, ο σκοπός της επιχειρησιακής αρχής είναι το να καθορίζει τις καθημερινές μας δραστηριότητες ώστε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε και για τις οποίες σας δώσω συγκεκριμένα, συγκεκριμένα παραδείγματα αμέσω. Γι' αυτό το τμήμα πάντως της διοίκησης να σας πω και δύο λόγια για τους χρήστες του ΣΑΤΣΕΝ. Έχουμε την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Εξωτική Υπηρεσία δράση. Αυτοί είναι οι κύριοι χρήστε της υπηρεσίας μας. Και α δώσω και κάποια παραδείγματα. Επίση οι χώρε μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Σάτσεν για να συμπληρώσουν ακριβώς τι δικέ τους δράσεις. Η Κομισιόν, τρίτε χώρε και διεθνείς οργανισμοί. Σήμερα το ΣΑΤΣΕΝ χρησιμοποιείται ως ένα πολιτικό διπλωματικό εργαλείο από τους, και από τους διεθνείς οργανισμούς όπως ε, ξέρω, διάφορες φύσεις πολιτικοί διεθνείς οργανισμοί. Να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι διεξοδικός ο κατάλογος, αλλά ενδεικτικός με επιχειρήσεις και αποστολές της Ένωσης. Με τη Γεωργία. Έχουμε ένα κέντρο μάλλον στη Γεωργία που ασχολείται ας πούμε με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, ε, στις ε, γειτονικέ περιοχές, ασχολούμαστε με το θέμα της μετανάστευσης, της πειρατείας, ε, κέρια σημεία της δραστηριότητας μας σήμερα με σημαντική βέβαια πολιτική σκοπιά και ασχολούμαστε και με άλλες χώρες, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα όπου έχουμε δραστηριότητες εκεί αλλά μας ενδιαφέρουν επίσης και οι θεομηνίες οι φυσικές καταστροφές οι ανθρώπινες καταστροφές Είμαστε πολιτική υπηρεσία, αλλά έχουμε κατά κάποιο τρόπο διπλού χαρακτήρα, διτού χαρακτήρα δραστηριότητες. Συμπληρώνουμε λοιπόν την ε, παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουμε τις ειδικές αποστολές εποπτείας και εποπτεύουμε επίσης και τη συμφωνία του Μίνσκ. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι συμφωνίες δεν εφαρμόζονται σωστά. Οπότε εμείς εντοπίζουμε τους τρόπους παρέμβασης σε απαγορευμένες περιοχές. Επίσης για την κατάσταση στη Συρία και με αυτή ασχολούμαστε. Παρακολουθούμε, ας πούμε, στην Λατάκια την τοποθέτηση στρατιωτικών ρωσικών μονάδων. Παρακολουθούμε την κίνηση αεροσκαφών, ελικοπτέρων. Υποδομή στρατιωτική, συστήματα εράμινας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ε, γενικότερα στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Και στην μετανάστευση επίσης έχουμε ρόλο και ιδιαίτερα παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης σε καθημερινή βάση για αυτά τα θέματα της μετανάστευσης. Παρακολουθούμε, ας πούμε, τις τουρκικές ακτές σε διάφορες τοποθεσίες ενδιαφέροντος και μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους δείκτες ώστε να έχουμε κάποια στοιχεία για να αξιολογήσουμε την εξέλιξη της μετανάστευσης. Παρακολουθούμε τους διακινητές όταν ανοίγονται στη θάλασσα και τις αφήξεις των μεταναστών με τα διάφορα πλωτά μέσα και στη θάλασσα λοιπόν που βλέπετε έχουμε έτσι μια σημαντική δραστηριότητα. Άλλη μια δραστηριότητά μας είναι η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής Βόρεια Κορέα συγκεκριμένα πυρηνικά όπλα και εμπροκειμένου προσπαθούμε να περιγράψουμε τις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, ποια μέσα αγκαθίστανται και τα διάφορα συστατικά αυτής της πυρηνικής δραστηριότητας. Ασχολούμαστε επίσης και με την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως στον Μπαγκλαντές. Και αυτός είναι και ο στόχος της δουλειά μας εκεί, ώστε να εξοργήσουμε την κατάσταση, να δούμε τι δραστηριότητες υπάρχουν από τους διάφορους φορείς, υποδομές, καταλήματα, ώστε να έχουμε μια όσο πιο ακριβή γίνεται της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Και τελευταίο συγκεκριμένο από το παράδειγμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα το πρωί είναι η πολιτιστική κληρονομιά που δεν είναι φυσική κατάσταση, μάλλον φυσική ιδιότητα αυτής της δραστηριότητα, αλλά στην περίπτωση του Ιράκ και της Συρίας, στη Μοσούλη στο Ιράκ συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε τα ερήπια μετά την καταστροφή από το ISIS μνημείων γιατί το ISIS ακριβώς χρησιμοποιούσε αρχαία για την χρηματοδότησή του Προσπαθούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση και τη μετακίνηση αυτών των αρχαίων. Προσπαθούμε λοιπόν να καταγράψουμε τα μνημεία πριν και μετά την καταστροφή τους και παρακολουθούμε την μεταφορά των διαφόρων κομματιών. Αυτά είναι λοιπόν τα συγκεκριμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων της Σάτσεν και να σας δώσω τώρα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τις δορυφορικές μας δραστηριότητες. Πράγματι τα τελευταία 8-10 χρόνια είδαμε μια τεράστια αύξηση στη δραστηριότητα της Άτσεν ακριβώς για να ανταποκριθεί στην γεωμετρική άνοδο πιθανών χρηστών των δραστηριοτήτων μας. Και από το 2013 έχουμε πολλαπλασιάσει τον αριθμό των προϊόντων μας επί τρία 2.200 προϊόντα παρακολούθησης παρήγαμε. Είχαμε και αύξηση των κατεβασμάτων των προϊόντων μας από τις χώρες μέλη. Αυτό υπερπολπλασιάστηκε, επί 20, 20 πλασιάστηκε η χρήση δηλαδή των δεδομένων των προϊόντων που παράγει το Σάτσεν από τις ε, χώρες μέλη. Να σας αναφέρω επίσης ότι πριν δύο χρόνια χρειάστηκε 30% της παραγωγής μας να το παραδώσουμε εντός 24 ώρου και σήμερα πάνω από το 75% αφού συλλεχθούν τα δεδομένα των προϊόντων μας παράγεται εντός 24 ώρου και κατεβάζεται λαμβάνεται δηλαδή ηλεκτρονικά συνεργασία. Έχουμε κάποια επίσημα έγγραφα που περιγράφουν ακριβώς την αποστολή μας και τις μορφές συνεργασίας με διάφορους εταίρους. Είναι τα επίσημα κείμενα τα οποία ακριβώς ε, προβλέπουν την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας και την αποφυγή των επικαλύψεων και βεβαίως προσπαθούμε να τηρήσουμε αυτούς τους κύριους προσανατολισμούς, πολιτικούς προσανατολισμούς και να προσφέρουμε υπηρεσίες προς τους πολίτες αλλά και τους διάφορους ενδιαφερόμενους και φορείς. Και να, επιτρέψτε μου να πω ότι όλες αυτές τις δραστηριότητες μας οδηγούν σε συγκεκριμένε εφαρμογές. Αυτό είναι βασικό και είναι σωστό να το ξέρουν οι πολίτες και οι φορολογόμενοι. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου για την διακυβέρνηση της υπηρεσίας μας και περιγράφει ακριβώς τους τρόπους συνεργασίας μας με την Κομισιόν και με άλλες υπηρεσίες, με τις χώρες μέλη και με παράγοντες εκτός Ένωσης. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό στη συνέχεια. Είχαμε την πρόσφατη πρόταση από την Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο για τη διευκόλυνση της νομοθεσίας ώστε να σε για να έχουμε περισσότερες συνέργειες στις δραστηριότητες μας ιδιαίτερα σε σχέση με το διαστημικό πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν σήμερα συμφωνίες με διάφορους εταίρους με το EDA, με τη Frontex στηρίζουμε την συνολική δραστηριότητα της Frontex μέσω διαφόρων τρόπων υποστήριξης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος επίσης και συγκεκριμένα να τονίσω μια πολύ συγκεκριμένη συνεργασία που έχουμε με το Κοπέρνικους που όπως ξέρετε ένα πρόγραμμα παρατήρησης με έξι κύρια στοιχεία κλίμα, θαλασσίες μεταφορές, ε, καταστάσεις εκτάξης ανάγκης κλπ. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Κοπέρνικους, με κονδύλια που προέρχονται από τον προπολογισμό της Ένωσης. Διεξάγουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες με το Κοπέρνικους και για το διάστημα εξετάζουμε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και για το δορυφορικό κέντρο προβλέπουμε ότι θα υπάρχει αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με την Κομισιόν και το Κοπέρνικος και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουμε κι εμείς στην εξέλιξη του Κοπέρνικους και της ασφαλείας του με τρόπο δυναμικό και ελπίζω στην εξέλιξη αυτή στις δραστηριότητες μας να ληφθεί υπόψη το ότι σε εμά εκπροσωπούνται πολλές χώρες μέλη και έχουμε επιστευτικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και ερχόμαστε σε επαφή με τους τελικούς χρήσες. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει η δικιά μας υπηρεσία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξέλιξη του Κοπέρνικους. Και καταλήγοντας, να σας δώσω ένα παράδειγμα των προϊόντων που παράγουμε στα πλαίσια του Κοπέρνικους. Έχουμε ενέρχικα προϊόντα, χάρτες αναχωρά, κατάσταση του δικοδικτύου, ζημιές και αποτίμηση, αποτίμησή τους, ε, ε, πολίτες ένωσης, ε, σύνορα κτλ. Και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στην εξέλιξη αυτού του χαρτοφυλακίου και χρειαζόμαστε επίσης την ανάδραση από τους χρήστες για να αναπτύξουμε αυτές τις υπηρεσίες μέσω του Κορπέρνικους με πιο ευαίσθητου χαρακτήρα προϊόντα ενδεχομένως στο μέλλον για να παρακολουθήσουμε και παράνομες δραστηριότητε και άλλα προϊόντα στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με τους χρήστες να αναπτύξουμε αυτή την υπηρεσία προς το Κοπέρνικους. Και δύο τελευταία στοιχεία το ΣΑΤΣΕΜ είναι μια γεωδορυφορική οντότητα. Γεωδορυφορική σημαίνει γεωγραφία και διάστημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο συνδυάζει τα δύο. Το γεγονό λοιπόν ότι υπάρχει μια θαυμάσια εξέλιξη της γεωδιαστημικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε όλο και πιο πολλούς δορυφόρους που βρίσκονται γύρω από την γη με, που συλλέγουν διάφορα δεδομένα ποικίλη ποιότητα. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε προσιλωμένοι στην εξέλιξη, γιατί συνέχεια μιλάμε για τα big data. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία ειστρέουν και θα πρέπει να έχουμε αυτοματοποιημένες δυνατότητες ανταπόκρισης στην αξιολόγηση αυτών των δεδομένων, παρέχοντας νέες υπηρεσίες έχοντας κατά νου ότι το δορυφορικό κέντρο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις χώρες μέλη της εξωτικής δράσης, τους μηχανικούς εταίρους και την Κομισιόν, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί από κοινού μια διαδραστική πλατφόρμα προς τους χρήστες, να έχουμε δηλαδή να παρέχουμε τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης χρήσης αυτής της πλατφόρμας με προϊόντα και δεδομένα τα οποία θα αποτελούν τον κατάλογο των προϊόντων μας, ο οποίος θα είναι πιο διαδραστικός. Αυτή είναι η αποστολή μας για το άμεσο μέλλον. Και τέλος, έχετε εδώ μια τελευταία διαφάνεια με την οποία ολοκληρώνω. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι σε εθνικό επίπεδο η συλλογή πληροφοριών είναι κάτι το κέρια σημασίας και ακόμα περισσότερο στην καθοδήγηση της υπηρεσίας κριτικής δράσης για την μετώπιση καταστάσεων όπως ε, τρομοκρατίας, μετανάστευσης, ε, περιφερειακών απειλών κλπ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι, ετοιμοπόλεμοι, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και βεβαίως να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές αλλού. Δεν μιλάω για τα εθνικά εργαλεία, αλλά για τα ευρωπαϊκά. Γιατί σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μεγάλη ικανότητα. Οπότε θα πρέπει εμείς ακριβώς να στηρίξουμε τις διάφορες δράσεις μας με ένα ελάχιστο, ελάχιστο ικανότητας συλλογής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα συζητάμε επειδή κάθε χρόνο πρέπει να συζητήσουμε τους πόρους του δορυφορικού κέντρου και επιτρέψτε μου να σας πω όχι τόσο διπλωματικά ότι κάθε χρόνο παλεύουμε και ζητιανεύουμε λίγες χιλιάδες ευρώ στα πλαίσια του ΠΔΠ 21-27 εκεί που γίνεται λόγος λαγή για δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ για άμυνα και ασφάλεια. 27 νομίζω για την 7 ετία. Μα συμπεριλαμβανομένων και των 13 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Άμυνας. 34 δις μάλιστα προτείνει η Κομισιόν Διαχείριση των Συνόρων Επίσης το εργαλείο άμυνας με τις αποστολέ, 10,5 δις. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των πόρων που αφορούν τις δομές συλλογή πληροφοριών και των υπολείπων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και ένα τελευταίο που έχω να πω αφορά τον αντίκτυπο του Brexit για το Σάτσερ που δεν είναι ουδέτερο για μας γιατί είναι ο δεύτερος δωρητής ή συνεισφέρον η Βρετανία στον προπολογισμό μας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ή όχι τελική συμφωνία για τον Brexit. Αν όχι, για μας θα σημάνει, αν δεν υπάρξει συμφωνία, μια μεγάλη έλλειψη πόρων και μείωση των δυνατοτήτων του δορυφορικού κέντρου. Και κάτι άλλο τελευταίο, σε σχέση με το Κοπέρνικους και το Σάτσεν. Αν δεν συμμετέχουμε δεόντω στο Κοπέρνικους, τότε πραγματικά θα δεχθούμε σοβαρό πλήμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό που είπατε το τελευταίο με απασχολεί πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το σημείο να περάσουμε στον κύριο Στασάν πριν ανοίξω τη συζήτηση που είναι υπεύθυνο πολιτικής ε, της μονάδας ε, ειδική ομάδας για το διάστημα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας. Έχετε το λόγο κύριε Στασάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εκ μέρους της κυρίας ε, Κάριν Κλάις ε, που είναι η ε, πρόεδρος της ειδικής αυτής ομάδας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και εμάς. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το Σάτσεν άρχισε τις δραστηριότητες της ανάλυσης ε, εικόνων παρατήρησης ήδη από το 1992 και από τότε, από τότε που άρχισε να ε, λειτουργεί συμμετείχε στην επιχειρησιακή υποστήριξη της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στην προηγούμενη και στην τωρινή μορφή της ε, είναι μοναδική, μοναδικό στο είδος του μπορεί να, χρησιμοποιεί, μπορεί να αξιοποιήσει ε, τις εικόνες και όλα τα στοιχεία να παρέχει πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μυστικής, μυστικών πληροφοριών και όπως ε, είπε και ο Διευθυντής ε, του ε, Δορυφορικού Κέντρου, η διακυβέρνησή του, διαχείρισή του είναι στα χέρια των κρατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιχειρησιακή κατεύθυνση βέβαια είναι ευθύνη του του διευθυντή. Γι' αυτό ακριβώς κάποια τεχνικά στοιχεία έχουν ε, ανατεθεί στην ειδική ομάδα ε, στην οποία συμμετέχω. Ε, η βάση δεδομένων έχει πολλές φορές αναθεωρηθεί το 2010, το 2018 Η απόφαση της λήψης αποφάσεων ε, για την ΚΕΠΑ και την ΚΠΑ ε, είναι τομεί τους οποίους βοηθά πολύ το δορυφορικό κέντρο, όλο και περισσότερο ε, βασιζόμαστε στο δορυφορικό κέντρο. Είναι ένα παράδειγμα συγκέντρωσης και άντλησης πόρων. Όλες όλοι οι οικονομικοί πόροι συγκεντρώνονται με συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της ύπαρξής του. Από πλευράς ε, ευρωπαϊκής προοπτικής πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας στρατηγικής όπως η υβριδικέ απειλές, η τρομοκρατία, η προστασία των συνόρων μεταξύ άλλων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται απαραίτητες ικανότητες για να, για να συνεισφέρει ε, στην ευρωπαϊκή αυτονομία. Γι' αυτό υπάρχει η Υπηρεσία Ασφαλείας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και υπάρχουν και πολλές συμφωνίες με τη Frontex. Από την άλλη, τώρα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο το πεδίο μάγης, έχουν ε, συντομευτεί οι χρόνοι σε ώρες αν όχι σε λεπτά. Ε, η άμεση διαθεσιμότητα εικόνων ήταν πάρα πολύ σημαντική για την επεξεργασία και την άντληση σημαντικών πληροφοριών και της δυνατότητας διάδοσης ε, με έγκαιρο και έγκυρο και ασφαλή τρόπο. Περνάμε λοιπόν από την παροχή προϊόντων σε μια συνεχή ροή πληροφοριών. Επίσης ενημερώνουμε ε, όλες τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα πληροφορικής. Υπάρχουν επιχειρησιακά και, επιχειρησιακές και τεχνολογικές προκλήσεις, ε, αλλά και διάφορα τεχνικά ζητήματα, γιατί οι σφορές των κρατών μελών δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ελάχιστη ήταν η αύξηση τον τελευταίο έτος. Ε, το αναπτυθέν κόστος από εισφορές σε τρίτους δεν επιτρέπουν την οικονομική σταθερότητα. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεισφέρει περισσότερο με το ε, επόμενο πι Υπάρχει και το ζήτημα του Brexit, όπως είπε ο Διευθυντής. Ε, υπάρχει περίπτωση μεγάλης μείωσης και στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών προτάθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2017 να υπάρχει μία διαβούλευση για το μέλλον του οργανισμού με σκοπό να εξετάσουμε τη μελλοντική κατάσταση του δορυφορικού κέντρου σε σχέση με τους σπόρους του. Ε, ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια τον Ιούνιο του 2018. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα με εναλλακτικές επιλογές και θα παρουσιαστεί μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2019 στα κράτη-μέλη. Περίπου 18 συμπεράσματα και συστάσεις συμφωνήθηκαν μεταξύ αυτών ότι το δορυφορικό κέντρο είναι πολύ σημαντικό για την ε, λήψη αποφάσεων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ε, και άμυνας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι μυστικές πληροφορίες, ε, οι ειδικέ πληροφορίες, πρέπει να βελτιωθούν αυξηθεί η συμμετοχή του δορυφορικού κέντρου σε αποστολές και επιχειρήσεις. Για να, πρέπει επίσης να βελτιωθεί η παρατήρηση γεωγραφική ε, ε, εικόνων και δορυφορικών εικόνων ε, και να είναι πιο κατάλληλες για διάδοση και να μεγιστοποιηθεί συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οργανισμούς της και τα κράτη-μέλη, όπως είπε ο Διευθυντής του και ειδικότερα στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. Το δορυφορικό κέντρο και η ειδική ομάδα για το διάστημα παραμένουν δεσμευμένοι σε αυτή την προσπάθεια και θα αρχίσουν συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για να ολοκληρώσω πρέπει να πω ότι το δορυφορικό κέντρο είναι ένα μοναδικό μέσο υποστήριξης ε, της ε, ε, ΚΕΠΑ. Υπάρχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις μπροστά μας και υπάρχει ανάγκη τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής συνεισφοράς τώρα διαμορφώνουμε ένα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον οργανισμό. Thank you very much. And, uh, thank you to... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. για τις ε, συνεισφορές σας. Ευχαριστούμε για την ε, πληροφόρηση. Και αρχικά θα θέλαμε να ε, ρωτήσουμε για τον ε, προϋπολογισμό. Όπως ε, τονίσατε και οι δύο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για το έργο σας και στο αβέβαιο περιβάλλον που βρισκόμαστε ιδιαίτερα στον όψη του Brexit. Θα ήθελα λοιπόν άμεσα ευθείαν να σας ρωτήσω ε, τι θα μπορούσαν, ποια θα μπορούσαν να ήταν τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα και επίσης αν έχετε ε, μία συγκεκριμένη παράκληση για εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσατε επίσης ε, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτήσατε γι' αυτό και αν θα μπορούσατε να το ε, να γίνετε πιο συγκεκριμένος για την επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ένα θέμα στο οποίο επιστρέφουμε ξανά και ξανά και αφορά την επικοινωνία Αναγνωρίζουμε την πρόκληση του προϋπολογισμού, όμως πάντοτε θα πρέπει να ε, πείσουμε τους πολίτες για ποιο λόγο υπάρχουν διάφορες ε, υπηρεσίες και αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας ε, σχετικά με τα όσα κάνετε και τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχετε Έχετε λοιπόν μια στρατηγική επικοινωνίας ευρύτερα. Επίσης αναφερθήκατε στο ότι έχετε μία ε, σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στην ΙΣΑ και ε, παρακαλώ ε, μπορείτε να μας πείτε για την σχέση της Σάτκεν με το, στο πλαίσιο αυτό. Και τέλος το Brexit, λέγοντας αρχής εξ αρχής ξεχαθάρα... καταλαβαίνετε ότι είμαι Βρετανίδα, αλλά μια Βρετανίδα που πιστεύει ότι το Brexit είναι ένα μεγάλο λάθος. Πώς ε, λοιπόν θα θέλατε να δείτε, να εξελίσσετε η μελλοντική σας σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτήν την πολύ κακή ιδέα. Και το τελικό μου ερώτημα. Το πρωί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για την τεχνητή νοημοσύνη και αναφερθήκατε ε, στο να μεταφερθούμε από το downloading στο συνεχόμενο feed. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, κάποιο στοιχείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τον προπολογισμό, το πρώτο σας ερώτημα, δεν ε, είναι το θέμα να πούμε θέλουμε περισσότερα χρήματα, οποιοδήποτε μπορεί να το πει αυτό πολύ εύκολα, αλλά το τι θα κάνουμε με, αυτές τις, με αυτά τα χρήματα, με αυτού τους πόρους. έχουμε να κάνουμε με χρήστες, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ζήτηση. Και ε, πάλι θα πρέπει να είμαστε δραστικοί, να παραμένουμε σχετικοί. Και για αυτό το πράγμα λοιπόν χρειάζεται να σκεφτούμε τις διάφορες πιθανότητες. Σύντομα έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο με τα 28 κράτη-μέλη μέσα Οκτωβρίου για να παρουσιάσω τις θέσεις μου ε, για το ε, όραμα μας ε, για την υπηρεσία για του χρόνου. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να βασίσουμε αυτή την ανάπτυξη σε τεχνολογικές λύσεις. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την τελευταία σας ερώτηση, περισσότερη αυτοματοποίηση στην υπηρεσία μας. Η ιδέα μου δεν είναι να πολυπλασιάσουμε τον αριθμό του προσωπικού, αλλά να έχουμε πιο αυτόματες ε, διαδικασίες και να χρησιμοποιήσουμε τις ορθές τεχνολογικές λύσεις να έχουμε μια ασφαλή πλατφόρμα που θα ε, δίνει πρόσβαση σε διάφορους ε, χρήστες. Και, δε, και γι' αυτό χρειάζεται όχι μόνο η υποδομή, αλλά ε, σε αυτή την πλατφόρμα να συνεισφέρουν διάφοροι εταίροι. Είπα ότι υπάρχει μια μεγάλη επανάσταση δεδομένων παραγόντων στον εμπορικό κόσμο, ενώ όπως είπε ο Νίκολας, έχουμε και κράτη-μέλη τα οποία κάνουν ε, προτάσεις ε, για πρόσβαση στα εθνικά του συστήματα. Και επίσης έχουμε τον δορυφόρο Κοπέρνικους ε, και θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να συλλέγουμε τα διάφορα δεδομένα, να έχουμε συμβόλαια με τους εμπορικούς παρόχους, θα υπάρχει κόστος ε, για αυτό και να έχουμε τα δεδομένα, τα εργαλεία ε, επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και βέβαια για όλο αυτό υπάρχει κόστος. Η προστιθέμενη αξία για τους τελικούς ε, χρήστες τώρα θα είναι εύκολη πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει μια κρίση, για παράδειγμα, μια καταστροφή θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να μπουν σε αυτήν την πλατφόρμα και να ε, συλλέξουν τα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για επίλυση της λύσης. Αυτή είναι η τεχνολογική προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε. Βέβαια, θα πρέπει να συνοδευτεί αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη, επανάσταση και με τις αναγκαίες δεξιότητες και το κατάλληλο προσωπικό δεν είναι βέβαια εύκολο να ε, προσλάβουμε το ανάγκαιο προσωπικό, θα πρέπει να είμαστε ελκυστικοί για να μπορέσουμε να βρούμε το αντίστοιχο προσωπικό. Επίσης όσον αφορά τους πόρους, ανέφερα την εξέλιξη του Κοπερνικούς στο πι δελτα πι μιλάμε για τη γραμμή του προϋπολογισμού που ανέρχεται στα 16 δις για την 7 η αυτή περίοδο το Κοπέρνικους ε, αντιστοιχεί σε 5 δις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ασφάλειας. Αυτό το οποίο δεν ανέφερα όμως είναι το γεγονός ότι το ε, ετήσιο εισόδημα της ε, ΣΑΤΣΕΝ είναι στα 26 εκατομμύρια. ετησίως και τα 50, το 50% προέρχεται από τις ε, άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών και 50% από την Επιτροπή, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό το πρόγραμμα Κοπέρνικους είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη υπηρεσιών ε, στο μέλλον. Αν λοιπόν με ρωτάτε πόσα εκατομμύρια ακόμα θέλω, θα ήθελα να σας πω ότι θέλουμε ότι η τεχνολογία και το Κοπέρνικους είναι σημαντικό, σημαντικά ζητήματα για αυτό. Επίσης έχουμε πρόσβαση σε έναν σε αυξανόμενη ποσότητα δεδομένα. Δεν έχουμε όμως τις τεχνικές δυνατότητες για να απορροφήσουμε αυτά τα δεδομένα. Όμως ε, τεράστια ποσότητα δεδομένων, δεδομένων είναι μια ευκαιρία διότι με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα και όσο περισσότερα δεδομένα τόσο πιο ωφέλιμο είναι για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι είναι δυνατόν να αναπτύξουμε μοντέλα και εργαλεία χρησιμοποιώντας αυτήν την ποσότητα δεδομένων και να έχουμε εύρωστες λίστες ε, στο τέλος ε, και στο ΣΑΤΚΙΑΝ έχουμε αρχίσει να αναπτύξουμε εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη για να έχουμε αυτόματο εντοπισμό στόχων, ε, το οποίο επίσης είναι χρήσιμο όσον αφορά την αυτοματοποίηση και την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, οι ψηφοφόροι, οι φορολογούμενοι θα πάνε τον Μάιο να ψηφίσουν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όλοι έχουμε την υποχρέωση να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο και ότι δεν σπαταλάμε πόρους αλλά τους χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σήμερα τα ε, έχουμε ε, τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν όλο και πιο πολύ τις υπηρεσίες του Σάκεν. Όπως είπατε υπάρχει μια στρατηγική επικοινωνίας ε, επειδή δαπανούμε τρομερή ενέργεια για να έρθουμε σε επαφή με τους χρήστες και τους πιθανούς χρήστες Υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο διοργανώνουμε τακτικά συναντήσεις, συνεδριάσεις ε, ε, στην υπηρεσία μας και η Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ θα μας επισκεφθεί μελλοντικά. Ε, εργαστήρια διοργανώνουμε για, για το Κοπέρνικους στο Παρίσι στις 11 Δεκεμβρίου και προσκαλούμε πολλούς χρήστες και πιθανούς ε, χρήστες να ακούσουν τις ιδέες μας ε, για την εξέλιξη των υπηρεσιών ε, και να, να απαντήσουμε στις ανησυχίες τους και τις επιθυμίες τους. Η στρατηγική επικοινωνίας λοιπόν είναι να επενδύσουμε σε τέτοια. Για παράδειγμα, χθε με κάλεσαν στην ΕΦΚΑ είναι άλλη μια υπηρεσία της ε, Επιτροπής ε, επίσης για να μιλήσω για πιθανές κοινέ δραστηριότητες στο μέλλον και βρισκόμαστε σε επαφή και με άλλες ε, υπηρεσίες για να δούμε πιθανότητα συνεργειών. Πηγαίνουμε στις διάφορες πρωτεύουσε για να συναντήσουμε τα κράτη-μέλη, να ακούσουμε τις ανάγκες τους, τις απόψεις τους. Ε, πιστεύω ότι κάλυψα λίγο πολύ τα διάφορα θέματα που αναφέρατε και φυσικά το πλαίσιο του διαστήματος είναι ένα πλαίσιο το οποίο μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, προσφέρει όλο και περισσότερες δυνατότητες και βέβαια ένα σημαντικός παράγοντας είναι η βιομηχανία, η ευρωπαϊκή βιομηχανία διότι η καινοτομία και οι εξελίξεις ε, έρχονται από τη βιομηχανία και αποτελεί συμφέρον μας να έχουμε στενή επαφή με τους βιομηχανικούς εταίρους, με τις startups, ε, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διότι έχουν λύσεις ε, για την χρήση αυτών των ε, δεδομένων. Και μπορούμε και επίσης εμείς να υποφεληθούμε. Και επίσης οργανώνουμε τις Industry Days, βιομηχανικές ημέρες, προσκαλούμε χρήστες από τα κράτη-μέλη, ε, υπηρεσίες ε, για να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να εξετάσουμε τις ε, λύσεις που έχουν οι εταίροι από την βιομηχανία και να παρουσιάσουμε και εμείς το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. που απαντήσατε ταυτόχρονα τόσες πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Στάση. Ευχαριστώ τον Πασκάλ για, την, για τις εκτενείς απαντήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τώρα τον ε, προϋπολογισμό, ε, ήταν ε, μια δύσκολη δράση είχαμε τα, τις ε, τρομοκρατικές απειλές, είχαμε αύξηση πέρσι και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με τα κράτη-μέλη, όμως ε, δεν θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που αντιμετωπίζει το ΣΑΤΣΕΝ. Τώρα θα αξιολογήσουμε όλες τις ε, δυνατότητες, όλα τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να συνεισφέρουν θα αξιολογήσουμε τον ε, μηχανισμό ανάκλησης κόστους, cost recovery mechanism, για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τα έσοδα, την σταθερότητα Τώρα όσον αφορά τα, την πρόσβαση στα κυβερνητικά συστήματα υπάρχει δυνατότητα για πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς χρέωση και όπως είπε ο Πασκάλ η συνεργασία με την Επιτροπή υπάρχει στο πλαίσιο του προγράμματος Κοπέρνικους και επίσης έχει γίνει πρόταση από την Επιτροπή να ενισχύσουμε αυτή τη συνεισφορά και σίγουρα θα εξετάσουμε αυτήν την ε, ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Όπως είπα, η χρονιά αυτή θα είναι σημαντική για την ε, συλλογή των ε, πληροφοριών. Τώρα όσον αφορά τα κράτη-μέλη θα έχουμε διάφορες δυνατότητες. Θα δούμε ποια είναι η πολιτική βούληση και πού μπορούμε να πάμε από εκεί. Όσον αφορά τους πολίτες τώρα, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Σατσέν είναι μια ιστορία επιτυχίας όσον αφορά την συλλογή και τη διαμονή, διανομή. Υπάρχει δυνατότητα ε, υποβολής ερωτήσεων για εθνικές ανησυχίες στον τομέα της ασφάλειας και το όφελος λοιπόν για τα κράτη-μέλη είναι τεράστιο. Οπότε ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Και φυσικά ε, η υπηρεσία μας είναι σημαντική και για την επιτύχηση της παγκόσμιας στρατηγικής και θα πρέπει να εφιστήσουμε περισσότερο την προσοχή στην σημασία αυτής της υπηρεσίας. Τώρα όσον αφορά το Brexit βέβαια είναι ένα θέμα όπως είπα είναι μια υπηρεσία ε, συλλογής πληροφοριών από τον ε, Μάρτιο του 19 αρκετοί θα χάσουν ε, την ε, πρόσβασή τους στην υπηρεσία θα υπάρξει μια οικονομική συνέπεια. Θα αποτελεί τρίτη χώρα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι για την ώρα ακολουθούμε μονάχα τις οδηγίες της Task Force 50. Επίσης, ε, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην ροή δεδομένων πληροφοριών που καταφτάνουν και να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση εγκαίρως στις πληροφορίες αυτές και φυσικά έχουμε την ε, μηχανική μάθηση που θα παίξει επίσης ρόλο σε αυτό. Είναι επίσης μια πρόσκληση και για την ύπατη εκπρόσωπο η οποία επιβλέπει τον, τις δραστηριότητες μας. Κάθε έργο το οποίο φτάνει στην υπηρεσία εξετάζεται αρχικά από την ε, ειδική tax force και αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι το εάν η, ε, το αίτημα αυτό ανταποκρίνεται σε ζητήματα κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, της ΚΕΠΑ σε αυτό ε, περιλαμβάνει και το πρόγραμμα Κοπέρνικους ε, και φυσικά θα πρέπει να αντιποκριθούμε ε, με τους πόρους που έχουμε. Όλα αυτά τα βήματα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για να έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου την προπιστοποίηση του χρήστη είναι μια μεγάλη πρόσκληση όλο και αυτό, όλο αυτό για μας και δεν θα πρέπει να επιβραδύνουμε την ε, διαδικασία και να αποφύγουμε ότι οι πληροφορίες φτάνουν πολύ αργά. Αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση λοιπόν για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, το εκτιμούμε ιδιαίτερος και που επίσης τονίσατε το σημαντικό έργο που κάνει η Σάτσεν, ιδιαίτερος ε, για τους ε, πολίτες. Και το έργο σας έμεσα ή άμεσα προστατεύει ε, αυτούς μας τους στόχους. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που ήρθατε σήμερα. Και έτσι ολοκληρώνουμε την πρωινή μας συνεδρία και θα συνεχίσουμε πάλι στις 2.30 το μεσημέρι.